przewodniczący! E, panie i panowie, koleżanki i koledzy, wznawiam posiedzenie. Άρχεται η συνεδρίαση, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα πρακτικά τη συνεδρίασης τη θεσινής ημέρα ε, εγκρίνονται και είναι στη διάθεσή σα. Έχετε παρατηρήσει, Δεν βλέπω ότι υπάρχουν παρατηρήσει, Κατά συνέπεια εγκρίνονται τα εν λόγω πρακτικά. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη που είναι η κοινή συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έκθεση των κυρίων Μπροκ και Φεχόφστατ για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αλλά και μια δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ακριβώς για το ίδιο θέμα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δηλαδή. Κυρία Αντιπρόεδρε και είπατε εκπρόσωπε, μόλις ξεκινήσαμε τις συζητήσεις μας. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μπρόκ για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ως εισηγητής και από την, υπηρεσία, από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επάτη, και Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτο σημαντικό βήμα για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Επιτευχθεί με τη Συμφωνία της Μαδρίτης. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι ακόμα αυτό οριστικό, διότι υπάρχει όλο το απαραίτητο περιθώριο χειρισμό για τη διαδικασία συναπόφασης, για το δημοσιονομικό κανονισμό των υπαλλήλων και τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και ε, τον οικονομικό προγραμματισμό, αλλά έτσι μπορούμε να προγραμματίσουμε τα επόμενα στάδια και ε, από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλουμε να τονίσουμε ότι την επιθυμούμε αυτή την υπηρεσία εξωτερική δράση. Ήταν επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλωστε, ήδη από τη συνταγματική συνέλευση να έχουμε έναν ύπατο εκπρόσωπο που θα συντονίζει τις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επιφορτίζεται με την ΚΕΠΑ την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία και θα έχει και στη διάθεσή του μια υπηρεσία που θα τον καθιστά ικανό ε, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απέναντι στο Συμβούλιο και απέναντι στον κόσμο όλο, ικανό να έχει μια θέση συνεκτική και να κάνει σωστά τη δουλειά του στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και να φροντίζει να μην είμαστε μόνο ένας παγκόσμιος πληρωτής αλλά και ένας παγκόσμιος πρωταγωνιστής. Όχι μόνο global payer λοιπόν αλλά και global player. Και νομίζω ότι είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Για μας σημαντικό ήταν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να έχουμε ως ύψιστο στόχο την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας ευθύς προς το κοινό συμφέρον των πολιτών της Ευρώπης, αλλά και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες να μην αλλάξουν τόσο πολύ, ώστε αυτό που έχει προκύψει ως κοινοτικό δίκαιο πλέον και ε, υπόκειται ε, στην κοινοτική ε, Ευρώπη να μην ξαναπέσει στην διακυβερνητική Ευρώπη και ε, στη συνεργασία των κρατών μεταξύ της. Νομίζω λοιπόν ότι καλά τα πήγαμε και επιτρέψτε μου ε, κύριε Επίτροπε ότι καμιά φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε περισσότερα πράγματα για τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Επιτροπή την ίδια. Θα ήθελα να πω επίσης αγαπητοί συνάδελφοι ότι στην αρχή υπήρξε κάποια διστακτικότητα, αλλά στη συνέχεια εμφανίστηκε πρόθυμο και το Συμβούλιο να ακούσει αυτά που είχε να πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να καταλάβει ότι το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα λόγου εδώ και συναπόφαση και για τον οικονομικό κανονισμό και ε, για ε, τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων. Γενικά έχουμε διαδικασία συναπόφασης και ήταν ε, σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε και έχουν γίνει και σε αυτό πρόοδοι. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από την εξασφάλιση της κοινοτική μεθόδου, να είμαστε βέβαιοι για την εξασφάλιση και των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου και τη διεύρυνση των ε, δικαιωμάτων του πάντα στα πλαίσια της συνθήκη Και αυτό όχι μόνο σε πολιτική εσωτερικών και ασφαλείας, και στην πολιτική εξωτερικών και ασφάλειας και στο μέλλον για πρώτη φορά θα ε, μας ρωτάνε και θα μας ενημερώνουν πριν ληφθούν οι αποφάσεις. Και όχι μόνο ακροάσεις, αλλά και πριν διοριστούν, ας πούμε, πρέσβεις. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε απόψεις και να ρωτάμε τους πρέσβεις πέρα από το δημοσιονομικό δικαίωμα που έχουμε, πέρα από το δικαίωμα που έχουμε να κυρώνουμε στο μέλλον συνθήκες με τρίτες χώρες και στην ενδιάμεση φάση θα έχουμε μια διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης εκ των προτέρων για να υπάρχει και μια κοινοβουλευτική διάσταση ε, στην εξωτερική πολιτική. Και ένα τελευταίο. Δεν θα κάνει το Κοινοβούλιο επιχειρησιακή εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι ε, αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας. Εμείς θέλουμε έλεγχο κοινοβουλευτικό και να μπορούμε να λέμε και όχι για σημαντικές αποφάσεις και για τον προπολογισμό. Να ελέγχουμε λοιπόν και γι' αυτό χρειαζόμαστε τα απαραίτητα εργαλεία και την ενημέρωση υπέρ των πολιτών, υπέρ του κοινοβουλευτισμού και νομίζω ότι έχουμε κάνει σημαντικό βήμα πρόοδο εδώ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Υπάτη εκπρόσωπο που τελικά κατάληξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπρόκ για τον λόγο σας. Καλό θα ήταν να είστε μέσα στο χρόνο σας όλοι. Σημαντικός ο λόγος, αλλά παρά τα αυτά προσπαθήστε να τηρήσετε τις προθεσμίες. Να καλωσορίσω και τον κύριο Σεύκοβιτς, ε, αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Καλώς ήλθατε κύριε Σεύκοβιτς ο Γκί Βερχόφσταντ ως εισηγητής. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Έλμαρ Μπρόκ και τον Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη που ήταν συνεισηγητές και διεξήγαγαν και τις διαπραγματεύσεις με την, με την κυρία Άστον και τις υπηρεσίες της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Η υπηρεσία δεν ξεκίνησε να λειτουργεί και πιστεύω αγαπητοί συνάδελφοι ότι μπορούμε να πούμε πως το αποτέλεσμα είναι ένα καλό αποτέλεσμα που μπορούν να υποστηρίξουν όλα τα όργανα και για την οποία μπορεί να είναι υπερήφανοι όλοι. Και μπορώ να επαναλάβω αυτά που είπε χτες ο Γάλλος Πρωθυπουργός ο κύριος Φιγιόν όταν δήλωσε ότι η υπηρεσία μπορεί να ξεπεράσει κάποια, ε, κάποιες κόκκινες γραμμές. Ε, να πω στον κύριο Φίγιο, αργήσατε. Η... Όταν ε, διαφωνήσαμε για την υπηρεσία, ξεπεράσαμε τις κόκκινες γραμμές της Γαλλίας. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, συνάδελφοι. Πρόκειται για πλήρη χρήση και ουσιαστική εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Κάτι τέτοιο προβλέπεται στη συνθήκη τη Λισαβόνα που ενέκρινε η Γαλλία να υπάρξει κοινή δραστηριότητα τη εξωτερική πολιτική στο μέλλον. Και αυτό που χρειαζόμαστε Πρόεδρε, δεν είναι μία μάχη οπισθοφυλακών για την, για την υπηρεσία, η οποία έχει αρχίσει, υπάρχει, αλλά τη σωστή χρησιμοποίησή της για να αναπτύξουμε μία πραγματικά ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Γιατί, α είμαστε ειλικρινεί, μέχρι τώρα δεν είχαμε μια πραγματική εξωτερική πολιτική τη Ένωση, ουδόλω. Θυμάμαι όταν ήμουν μέλο του Συμβουλίου του 2002, είχαμε δαπανίσει 50 δευτερόλεπτα για τον πόλεμο στο Ιράκ, που ήταν το μεγαλύτερο θέμα εξωτερικής πολιτικής εκείνη την εποχή. Την εποχή εκείνη η Ευρώπη δεν ήταν ικανή να συζητήσει καν, όχι να αποκτήσει κοινή θέση το ζήτημα. Δεν μπορεί να επαναληφθεί κάτι τέτοιο, όχι σε αυτόν τον πολυπολικό κόσμο της σήμερα. Δεν είναι επιλογή, δεν είναι, δεν, δεν, δεν είναι ουσιαστική δυνατότητα αυτή. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα η κυρία Άστον είναι αυτή που θα πρέπει να αναλάβει την ε, δράση. Και το μήνυμά μας είναι η υπηρεσία θα χρειαστεί σαφή καθοδήγηση, σαφή ηγεσία. Και η συνθήκη κυρία Άστον σας έδωσε πολλές εξουσίες για να κάνετε κάτι τέτοιο. Έχετε το δικαίωμα να συγκαλείτε Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών ακόμα και με βραχυπρόθεσμη πρόσκληση. Έχετε τη δυνατότητα να λάβετε πρωτοβουλίε γιατί είσαστε αντιπρόεδρο τη Επιτροπή. Έχετε επίση την ευθύνη να παρέχετε τις γενικές καθηγητήριε γραμμές για τα στρατηγικά συμφέροντα τη Ένωση και όλε οι ευθύνε αυτέ υπάγονται στις δικές σας αρμοδιότητες και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών σας. Μία συμβουλή επιτρέψτε μου να σας δώσω μόνο στο τέλος όλων αυτών των διαπραγματεύσεων μαζί σας. Αναπτύξτε την υπηρεσία σαν κοινοτικό εργαλείο. Η επιτυχία της Ένωσης χτίστηκε στην κοινοτική προσέγγιση, στην κοινοτική μέθοδο. Μόνο όταν χρησιμοποιούσαμε, χρησιμοποίησαμε την κοινοτική μέθοδο, προχωρήσαμε και πετύχαμε. Δείτε την ενιαία αγορά. Όπου κάτι τέτοιο δεν χρησιμοποιήθηκε, είχαμε στασιμότητα, υποχωρητικότητα. Πώς η Ένωση, για παράδειγμα, απάντησε στην οικονομική κρίση. Μόνο λοιπόν μέσω της μεθόδου αυτής μπορούμε να πετύχουμε. Και πραγματικά μέσω της διαμόρφωσης πραγματικών συμφερόντων της Ένωσης χωρίς παρέμβαση των κρατών μελών που θα μπορέσετε να προχωρήσετε μια εξωτερική πολιτική της Ένωσης και τούτο θα γίνει χρησιμοποιώντας τα προσόντα και την εμπειρογνωσύνη που έχετε στη διάθεσή σας για να μπορέσετε να εντοπίσετε αυτή, τι, αυτά τα συμφέροντα. Και βεβαίως εσείς θα έχετε και την ευθύνη να προασπίσετε τα συμφέροντα της Ένωσης. Διότι κατά την άποψή μου και κατά την άποψη του Κοινοβουλίου αυτό είναι, που είναι καλό για την Ένωση είναι καλό και για τα κράτη-μέλη και άρα καλό και για τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε η κυρία Άστον έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μεταξύ σα για να συζητήσω ένα από τα σημαντικότερα θέματα τη Ευρωπαϊκή Ατζέντα, τη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής δράση. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω ευγνωμοσύνη για τον τρόπο που συντάχθηκαν μαζί μου οι εισηγητέ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κύριος Μπρόκ, ο κύριος Φερχόφστατ και ο κύριος Γκουαλτιέρη. Επίση, η ΑΦΕΤ, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, η Επιτροπή Γιούρι και η Επιτροπή ε, Οικονομικών Υποθέσεων. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταφέραμε πάρα, πολύ, πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες και φτάσαμε σε ένα κοινό πλαίσιο εργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σεύκοβιτς, την ε, Ισπανική Προεδρία υπό τον Μιγγέλ Μαρτίνεφ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις νομικές υπηρεσίες οι οποίες μας υποστήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ήρθε ο χρόνος να αποφασίσουμε, αγαπητά μέλη. Τα πρόσφατα, τους πρόσφατους μήνες έγινε μεγάλη συζήτηση για τα διαδικαστικά και διοικητικά θέματα. Η, τα θεμέλια είναι ένας βασικός ε, σκοπός και Υπάρχουν πολλοί λόγοι, πληθώρα λόγων για τη σύσταση αυτής της υπηρεσίας, γιατί ήρθα σε επαφή με κυβερνήσεις, με στρατιωτικές αποστολές και με αντιπροσωπείες ανά τον κόσμο. Πριν μπω στις λεπτομέρειες, θα ήθελα να σας πω κάτι για το όραμα αυτής της υπηρεσίας ως προς το μέλλον. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή και ο καλύτερος τόπος να θυμηθούμε γιατί η υπηρεσία είναι τόσο σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αποτελεί μία μεγάλη αλλαγή μέσα στα πλαίσια των γεωπολιτικών δεδομένων. Δεν μπορούμε να δρούμε διαφορετικά τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με έναν κόσμο που ολοένα και εξελίσσεται. Θα πρέπει να, να προωθήσουμε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πιο συνεκτικό τρόπο και θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν πληθώρα μέσων και πόρων, ε, σχέσεων και πραγματογνωμοσύνης για να μας βοηθήσουν για έναν σταθερό κόσμο. Τώρα θα πρέπει να συμβάλλουμε με όλα αυτά τα στοιχεία έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε την επίδρασή μας, ιδιαίτερα σε μέρη του κόσμου όπου υπάρχουν μεγάλοι κλειδονισμοί. Από την Γάζα, στην Αϊτή, στην Ανατολική Αφρική, στα Βαλκάνια, αυτά είναι τα συμπεράσματά μου. Η εξωτερική δράση αφορά διάφορες επιμέρους πολιτικές και βεβαίως η διπλωματία δρά διαφορετικά αν πρόκειται για διαχείριση κρίσεων ή ανθρωπιστική βοήθεια. Και πολλοί συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να συμβάλλουν. Θα ήθελα να τιμήσω τους συναδέλφους και νομίζω ότι μπορούμε να δράσουμε από κοινού μέσω μιας κοινή πολιτικής στρατηγικής. Η φιλοδοξία μετατρέπεται τώρα σε πραγματικότητα. Πιστεύω ότι όταν μιλάμε θα εισακουόμεθα και όταν αναλαμβάνουμε δράση, η δράση μας θα οδηγήσει σε μεγάλες διαφορές. Μιλάμε για ευάλωτα, ευάλωτες χώρες, παράνομη μετανάστευση ε, και πιστεύω ότι αν, αν δράσουμε από κοινού θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, δηλαδή τη διπλωματία, την πολιτική δέσμευση, την ε, ανταπόκριση σε στρατιωτικά, ε, σε στρατιωτικά δεδομένα και δράσεις έτσι ώστε να προωθήσουμε την σταθερότητα και την ειρήνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου. Είδα τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν δρούμε από ε, κοινού. Είδα τι καταφέραμε με την Αταλάντα στην Ανατολική Αφρική, αλλά είδα ότι μπορούμε και ε, επιγείως να δράσουμε. Δηλαδή, οι στρατιωτικές μας αποστολές βοήθησαν πάρα πολύ και πιστεύω για να επιληθούν τα θέματα θαλάσσης θα πρέπει να δράσουμε επί ξηράς. Ο κύριος Πίγμπαλξ ακριβώς τόνισε, αυτό τόνισε. Και όταν ήρθαμε σε επαφή με τους επικεφαλείς των κρατών της Αφρικής, Μοζαμβίκης, Σεϊχελών, Κένιας και Τανζανίας είδαμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε επιτοπίως για να βρούμε λύσεις και για να υποστηρίξουμε τη Σομαλία ώστε να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Ξέρω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά για το μέλλον. Είμαι ιδιαίτερα φιλόδοξη, το ομολογώ, διότι πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να κινηθούμε προς τα μπρο, να λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία. Έχουμε μια καλή συμφωνία επιτάπητο, μια ε, σειρά δηλώσεων και μια, ένα σχέδιο απόφασης. Τα υποβάλλω σήμερα στις διαδικασίες σας. Θα ήθελα να τονίσω ορισμένα ειδικά σημεία για το πώς μπορούμε να βρούμε τις σωστές δικλείδες ασφαλείας που είναι σημαντικές για αυτό το σώμα. Καταρχήν, το κείμενο καθιστά σαφές ότι διασφαλίζουμε την κοινωνική μέθοδο εκεί όπου υπάρχει. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα συνεργαστεί με τις υπηρεσίες της ε, Επιτροπής ως αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ξέρω ότι το θέμα της πολιτικής λογοδοσίας είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι βρήκαμε ένα πολύ καλό πλαίσιο μέσω των πολιτικών ε, δηλώσεων ω προς την πολιτική λογοδοσία. Αναμένω στην ανταλλαγή πληροφοριών με την ανταλλαγή πληροφοριών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι συνεργάτες μου δίνουν, προσδίδουν μεγάλη σημασία σε αυτή την ε, πτυχή του θέματος. Δεν θα μπορέσω να είμαι παρούσα όπως θα ήθελα στις συζητήσεις σας ε, εξαιτίας των ε, καθηκόντων μου. Όμως θα προσέρχονται άλλοι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, επίσης θα λογοδοτεί η Τρόικα ή εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Ως προς τη λογοδοσία υπάρχουν εγγυήσει έτσι ώστε να υπάρχει μια σωστή, μια χρηστή δημοσιονομική διαδικασία ως προς τις απαλλαγές μέχρι τις ε, εξουσίες περί προϋπολογισμού και τις αντιπροσωπείες. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή διαχειριστική ομάδα μέσα στα πλαίσια μιας γενικής γραμματείας και έναν επικεφαλής στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Διοίκησης. Επίσης, έχουμε συγκεκριμένη αναπτυξιακή πολιτική και μέσα, διότι δεν πρέπει να χάσουμε από τον ορίζοντα την αναπτυξιακή μας πολιτική. Η αναπτυξιακή πολιτική είναι ύψης της σημασίας για την εξωτερική μας δράση μας προβάλλει στο ε, διεθνές παρασκήνιο ως βασικό δωρητή. Γι' αυτό αυτό, αυτό το σκέλος έχει σημασία και στις ε, διμερείς μας σχέσεις. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να αποσπαστεί από την εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό δημιουργούμε μια μεγάλη κοινή πλατφόρμα για να συνεργαστούμε full και υποφαινόμενοι θα συνεργαστούμε έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και να προωθήσουμε τους αναπτυξιακούς στόχους. Πέμπτον, έχουμε μία εξισορροπημένη συμφωνία ως προς το προσωπικό γιατί τα κράτη-μέλη θέλουν τουλάχιστον να πλαισιώσουν το 1 τρίτον του προσωπικού από εθνικούς διπλωμάτες, ενώ παράλληλα θα πρέπει το 60% να είναι μόνιμο προσωπικό. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ίση γεωγραφική κατανομή και ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων. Είμαι ε, υπέρ αυτού. Θα πρέπει η υπηρεσία αυτή να αντικατοπτρίζει τη διαφορετικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι καλύτεροι διπλωμάτες θα φέρουν στην υπηρεσία την πολυγλωσία. Έκτον, θα είδατε την ε, δήλωσή μου για την κεντρική διοίκηση της ΕΙΕΒ. Θα πρέπει να έχουμε μια κοινή κατανόηση για την εικόνα της υπηρεσίας. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει τα πράγματα να τεθούν σε σωστή βάση και μετά να γίνουν οι αναθεωρήσεις ανάλογα με τις εξελίξεις μου υποβάλατε πολλές ερωτήσεις για την οικοδόμηση της ειρήνης και τη διαχείριση της κρίσης. Θα ασχοληθούμε με τον προγραμματισμό και την ανταπόκριση σε κρίσεις, σε κατάσταση κρίσεως καθώς και οικοδόμηση της ειρήνης. Θα συνεργαστούμε σε στενή συνεργασία υπό τη δική μου άμεση ευθύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω τον διακυβερνητικό χαρακτήρα αυτών των πολιτικών. Θα πρέπει να συντονιστούν οι δραστηριότητες των διαφόρων τμήματων της ΕΕ και θα πρέπει να υπάρξει πλήρης συντονισμός μεταξύ όλων των υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε σχέση με την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την ε, ιδιαίτερη φύση του κάθε τμήματος. Επίσης, θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ειδικών εκπροσώπων και των επιμέρους τμήματων της υπηρεσίας. Επίσης, έχουμε προσδώσει μεγάλη σημασία πάντα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μια προτεραιότητα που συμμερίζομαι και υπόσχομαι ως ύποτη εκπρόσωπος ότι θα προωθήσω τα ανθρώπινα δικαιώματα και την χρηστή διακυβέρνηση ανά τον κόσμο έτσι ώστε να διέπουν κάθε επιμέρους τμήμα της πολιτικής μας. Αυτό σε επίπεδο κεντρικής εκπροσώπησης και σε επίπεδο αντιπροσωπιών. Πιστεύω ότι έτσι θα προωθήσουμε τους στόχους μας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης για να προωθήσουμε την εξωτερική μας πολιτική. Χρειαζόμαστε μια κοινή πλατφόρμα για να προωθήσουμε τα επιμέρους προγράμματά μας. Θα πρέπει να έχουμε τα μέσα και τους σωστούς ανθρώπους για να αρχίσουμε με την πραγματική εργασία. Συμφωνώ με τα όσα προτάθηκαν από τα μέλη και θα τα προωθήσω στο Συμβούλιο. Επίσης, έχει προταθεί ένας προϋπολογισμός και ένας τροποποιητικός προϋπολογισμός για το 2010. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και πιστεύω ότι η αυριανή ψηφοφορία είναι ένα ιστορικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να πραγματοποιήσουμε αυτό το κοινό όραμα για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Thank you, Madam Vice President. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε και είπατε εκπρόσωπε. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Σεύκοβιτς, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, κύριε, είπατε εκπρόσωπε αγαπητή κάθε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την γνωμοδότηση και να υποστηρίξω την ε, υιοθέτησή του. Θεωρώ ότι η ψηφοφορία αυτή θα είναι μια σημαντική στιγμή για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και ένα σαφές μήνυμα ότι η νέα υπηρεσία λαμβάνει την δημοκρατική υποστήριξή του σώματό σα, κάτι πολύ σημαντικό. Η απόφαση αυτή θα είναι και η σωστή, και η σωστή ε, παρουσίαση των συζητήσεων για την εξωτερική δραστηριότητα της Ένωσης. Και πρέπει να εκφράσω την ιδιαίτερη εκτίμησή μου για την ε, έντονη δραστηριότητα της κυρίας Άστον ως είπα της εκπροσώπου του τελευταίους μήνες. Δεν δημιουργούμε κάθε μέρα και μια υπηρεσία. Κάθε μέρα ήταν δύσκολη, περίπλοκη, πέτυχε όμως μέσα σε 7 μήνες να ε, δημιουργήσει αυτή την πολιτική συνένεση, σε 7 μήνες από το, τη θέση ισχύ της νέας συνθήκης, κάτι πολύ σημαντικό. Και τούτο νομίζω αποδεικνύει ότι η κάθε άστον πέτυχε μια σωστή εξισορρόπηση των ε, προτάσεων που είχε θέσει στο ξεκίνημα. Η απόφαση ωστόσο όπως διαμορφώθηκε έπρεπε να περάσει από την διαδικασία δημοκρατικού ελέγχου, μια διαδικασία που νομίζω ότι ήταν θετική στον τετραμερή διάλογο με τον κύριο Μωρατίνος και μέλη του Κοινοβουλίου ε, τους συζητητές Μπροκ, Φεχόφστατ και Γκουαλτιέρη και με μένα προσωπώντας την Επιτροπή μπορώ να σας πω ότι ε, Ψάξαμε κάθε διάταξη, κάθε άρθρο, προσπαθώντας να βρούμε την βέλτιστη δυνατή λύση. Και πιστεύω ότι το πετύχαμε. Η συζήτηση έμεινε, στάθηκε σε τρεις τομείς. Πρώτον, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η υπηρεσία θα είναι απόλυτα τμήμα του ευρωπαϊκού συστήματος. Το πετύχαμε νομίζω, θα έχουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Δεύτερον, πώς θα εξασφαλίσουμε σωστή οικονομική και χρηματοοικονομική λογοδοσία. Και εδώ εξετάσαμε όλες τις δυνατότητες και είμαι βέβαιος ότι παρότι δημιουργούμε κάτι νέο, οι πόροι θα, το σύστημα θα περιλαμβάνει όλους τους σωστούς, ε, τις σωστές δικλείδες λογοδοσίας. Τρίτο σημείο συζήτησης, αναπτυξιακή βοήθεια πώς μπορούμε να διαχειριστούμε όσο καλύτερα γίνεται κρατώντας το κοινοτικό πνεύμα και εξασφαλίζοντα, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα δημοκρατικού ελέγχου του Κοινοβουλίου. Και εδώ ε, το σκεφτήκαμε, το ξανασκεφτήκαμε, βρήκαμε δημιουργικές λύσεις και εν τέλει νομίζω παρέχουμε ένα κείμενο που επιτρέπει τις καλύτερες δυνατές συνέργειες με εμπειρογνωμοσύνη από τα κράτη-μέλη, από την Επιτροπή την επιτόπια εμπειρογνωμοσύνη των αντιπροσωπιών μας, επιτρέποντας έτσι να έχουμε μια πραγματικά αποτελεσματική παρουσία της Ευρώπης προς τα έξω. Περιμένω την υποστήριξη της η Επιτροπή στην απόφαση αυτή μέσα στο μήνα. Είμαστε σίγουροι, είμαι σίγουρος ότι και η Επιτροπή θα συνεργαστεί με την ύπατη εκπρόσωπο, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία στις τελικές της φάσεις και να περάσει και η δημοσιονομική διαδικασία ώστε να έχουμε και πραγματικά να έχουμε μια εξαιρετική δουλειά για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ήδη από φέτος. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Επιτροπή Ανάπτυξης. Το λόγο έχει ο κ. Κάσμαρεκ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Είπατη, εκπρόσωπε, κύριε Επίτροπε, κύριε και κύριοι, καλό το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Το κείμενο είναι καλύτερο από το αρχικό. Θα ήθελα να δηλώσω τις δικές μας προθέσεις. Εμείς τι θέλαμε. Καταρχάς να επικεντρωθούμε στους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής και να λαμβάνονται αυτή η υπόψη σε πολλούς τομείς πολιτικής. Με άλλα λόγια, δεν επιθυμούμε η αναπτυξιακή πολιτική να αποτελεί αποκλειστικά ε, και μόνο ένα κλάδο ε, που να είναι εξάρτητος από όλους τους άλλους. Υπάρχει Επίτροπος Ανάπτυξης που θα πρέπει να συνεργάζεται με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και να μην εκπροσωπείται η Ένωση μόνο από επαγγελματίες διπλωμάτες, αλλά και από πρόσωπα που ασχολούνται με την αναπτυξιακή βοήθεια, με το εμπόριο και με ε, άλλα. Κύριος Ιβο Στρέιτσεκ. Πάνε, πάνε Κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, κύριε Επίτροπη, κύριε Αντιπρόεδρε, πιστεύω ότι το κείμενο στο οποίο φτάσαμε είναι ένα συμβιβασμός και όπως όλοι οι συμβιβασμοί έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Αυτό που είναι θετικό είναι ότι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να λογοδοτήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με, τη, με θέματα πολιτικής και δημοσιονομικής λογοδοσίας. Θα πρέπει όμως να ενισχυθεί αυτή η τάση έτσι ώστε να συμβαδίζει με θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ως ε, προς την ε, πρακτική λειτουργία, είναι κρίμα διότι η έκθεση δεν αντικατοπτρίζει τη δική μας γνώμη που υποστήριξε και το ΕΛΚ και οι φιλελεύθεροι. Θα θέλαμε να αποσαφηνίσουμε τις ευθύνες και αρμοδιότητες, ιδιαίτερα ως προς τον Γενικό Γραμματέα, δυνάμει του άρθρου 207 και 208 της Συνθήκης. Ο κύριος Γκουαλτιέρη έχει το λόγο από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Ήπατη, εκπρόσωπε. Κύριοι Αντιπρόεδρε. Αυτή η έκθεση δεν είναι μια απλή γνωμοδότηση, αλλά ε, είναι απότοκη μιας ε, κοινή εργασίας και μιας κοινή διαπραγμάτευσης και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ισπανική Προεδρία και την ύπατη εκπρόσωπο. Το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο για να βελτιώσει το κείμενο της απόφασης που θα πρέπει να εγκρίνει το Συμβούλιο. Η συμφωνία και ο συμβιβασμός της Μαδρίτης μας οδήγησαν σε ένα ενωτικό αποτέλεσμα με βάση τη συνεισφορά Μπροκ Φερχόφστατ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορούμε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα της πολιτικής μας ως προς τη, με την ύπαρξη μάλλον μιας εξωτερικής υπηρεσίας και πιστεύω ότι θα υπάρχει πλήρης δημοκρατικός έλεγχος από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν πρέπει να υπερβούμε. Και ακριβώς επειδή μπορέσαμε να ασκήσουμε πλήρως ε, τα, τις εξουσίες και τα προνόμια μας με βάση αυτές τις κόκκινες γραμμές και την ενδεχόμενη υπέρβασή τους θα υπάρχει μια πιο δημοκρατική και ευρωπαϊκή υπηρεσία η οποία θα οδηγήσει σε μια συνεπή πολιτική ως προς την εξωτερική μας δράση χωρίς να υποσκάπτει τις αυτόνομες πολιτικές ή την ευθύνη της Επιτροπής. Αυτό έχει μεγάλη σημασία ως προς τα προνόμια, ε, νομοθετικά προνόμια και δημοσιονομικά ιδιαίτερα κατά τους επόμενους μήνες για να ορίσουμε τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και το δημοσιονομικό κανονισμό όπως ορίζει αυτό το κείμενο και για να εποπτεύσουμε ως προς τον τρόπο στελέχωσης της υπηρεσίας για να τηρήσουμε το γράμμα και το πνεύμα της Συμφωνίας της Μαδρίτης, έτσι ώστε να εκπροσωπείται και το προσωπικό μέχρι την κορυφή της υπηρεσίας μέσα στα πλαίσια μιας υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής και θα υποστηρίξουμε πλήρως αυτό το σχήμα διότι είμαστε υπέρ της κοινοτικοποίησης της εξωτερικής μας πολιτικής που προβάλλει και η Συμφωνία της Μαδρίτης. Ο κύριος δεν δεν είναι εδώ από ό,τι βλέπω. Η κυρία Λούνατσεκ έχει το λόγο για την Επιτροπή Γυναικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Άστον, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι. Τώρα έχω διπλή ιδιότητα. Μιλώ και ε, ω εισηγήτρια τη Επιτροπή Γυναικών, αλλά και ω κοιόδη εισηγήτρια των Πρασίνων. Και τα δύο εκπροσωπώντα τη συνάδελφό μου, Φρανσίσκα Μπράτμερ που γέννησε ένα κοριτσάκι πριν από 1,5 μήνα και ανέλαβα εγώ την εργασία αυτή. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω και να την υποστηρίξω για αυτή τη δουλειά της. Η Επιτροπή Γυναικών έχει θέσει το κέντρο βάρου στο εξή ζήτημα. Η ισότητα των φύλων ε, θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και στη σύνθεση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Το καταφέραμε αυτό, είσαι εκπροσώπηση περίπου ανδρών και γυναικών και ελπίζω κυρία Άστον και ε, στη συνεργασία σας και θεωρώ ότι η ισότητα των ευκαιριών θα γίνει σεβαστή. Στο άρθρο 157 της συνθήκης ορίζει πώς ε, ρυθμίζονται όλα αυτά, θα πρέπει να γίνουν και πραγματικότητα. Και στην επιλογή του προσωπικού σας να βεβαιωθείτε ότι θα έχετε εκπροσώπηση γυναικών σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδο ε, κεφαλής αντιπροσωπείας. Ως και ηγήτρια των Πρασίνων τώρα θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Μπρόκ, τον κύριο Φερχόφστατ και τον κύριο Γκουαλτιέρη και να του ευχαριστήσω για την συνεργασία και να πω ότι από κοινού καταφέραμε να περάσουμε πολλέ βελτιώσει σε σχέση με το αρχικό κείμενο για μια εξωτερική πολιτική πιο συνεκτική, πιο αποτελεσματική, κοινή σε τελική ανάλυση. Εξού και υποστηρίζει η πολιτική μου ομάδα τη σημερινή έκθεση και αύριο θα την υπερψηφίσουμε μια ισχυρή δομή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την αναπτυξιακή πολιτική. Μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο θέλουμε. Και θα έχουμε οι μέλλοντε πρέσβει τη Ένωση, ανδρών και γυναικών, θα πρέπει να έρχονται να κάνουν ακρόαση εδώ πριν αναλάβουν. Και επίση να έχουμε και ένα διαφανή ε, προπολογισμό για την εξωτερική πολιτική. Ε, λίγο μετριάζεται ο ενθουσιασμό μα, διότι δεν υπάρχουν σαφεί δομέ για την πολιτική ε, πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων και δεν έχουμε σχεδόν καθόλου προξενικές υπηρεσίες για τους πολίτες της Ένωσης στη νέα αυτή υπηρεσία. Θέλουμε λοιπόν επίλυση ε, των διαφορών με ειρηνικό τρόπο, με πολιτικό τρόπο. Ε, ο συμβιβασμό που προέκυψε δεν μας ικανοποιεί 100% αλλά με καλή βούληση Κυρία μπορούν αυτά να εφαρμοστούν, αλλά η φιλοδοξία σας να πάει και προς την κατεύθυνση ε, περιορισμού εθνικών συμφερόντων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, τον προεξάρχοντα ρόλο του στρατού, όπως έχει δείξει η Γαλλία το τελευταίο διάστημα. Τελειώνω. Ε, κοινή ευρωπαϊκή δράση λοιπόν και κοινή ευρωπαϊκή νοοτροπία με υποστήριξη του Κοινοβουλίου και όχι τόσο πολύ των κρατών μελών. Ευχαριστούμε σας είπα. Παρακαλώ συνάδελφοι. Ε, από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ήρθε ο κ. Σκάλφιν και του δίνω το λόγο. Πρόεδρε, κυρία Άστον, ένα από τα σημαντικότερα θέματα που τέθηκαν τους τελευταίους μήνες ήταν το ενδεχόμενο να έχει το, η δυνατότητα, η υποχρέωση μάλλον να δοθεί στο Κοινοβούλιο η πραγματική αρμοδιότητα ε, κρίσης και απόφασης για τις, εξωτερι, για ε, δαπάνες για, τις για την εξωτερική υπηρεσία της Ένωσης. Ε, τέθηκαν πολλά ερωτήματα για τη διαφάνεια και την ε, ε, λογοδοσία και χαίρομαι που κατορθώσαμε να βρούμε τις ε, βέλτιστες απαντήσεις για να μπορέσει να επιτρέψει την υιοθέτηση ενό ψηφίσματο από το Κοινοβούλιο. Οι σαφείς απαντήσει για τη δημοσιονομική διαδικασία μα επιτρέπουν να πιστεύουμε ότι η πολιτική θα υλοποιείται από όλα τα εμπλεκόμενα όργανα. Προσπαθήσαμε να μην καθυστερήσουμε την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να δείξουμε ότι οι μηχανισμοί που, που εισάγονται λειτουργούν πλήρως και προς όφελος των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, λέει ο κύριο Μάωρο. Αυτό που γίνεται κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο είναι αυτό που καθιστά πιο συγκεκριμένη την ανάγκη να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό η Ευρωπαϊκή Διπλωματική Υπηρεσία. Η επίτευξη αυτής της πολιτικής συμφωνίας θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα άριστο σημείο ως ένα άριστο ξεκίνημα και ως ένα θετικό μήνυμα για την ουσιαστική λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Οι στόχοι που εντοπίσαμε, να είναι μια ισχυρή υπηρεσία δηλαδή, να επιτρέπει στην Ένωση να ενισχύσει το ρόλο της στην διεθνή σκηνή, η σπουδαιότητα της διαφύλαξης και ενίσχυσης της κοινωνικής μεθόδου στην ίδια την υπηρεσία και η εξασφάλιση ελέγχου πολι πολιτικού ελέγχου και δημοσιονομικού ελέγχου από το Κοινοβούλιο θα εξασφαλίσουν, είμαι πεπισμένο απτά αποτελέσματα. Παραμένουν ωστόσο εκρεμεί κάποια ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν και που είναι αποφασιστικά για την υλοποίηση τη Υπηρεσία. Μιλώ για την αμφιλεγόμενη στάση πολλών κυβερνήσεων. Οι κόκκινε γραμμέ που ανέφερε ο συνάδελφο κ. Γκουαλτιέρη, έστω κι αν ε, παραβιάστηκαν στην πρόσφατη συμφωνία της Μαδρίτης, βαρύνουν πάντως άτυπα δεδομένης ακριβώς της επαμφωτερίζουσα θέσης πολλών κυβερνήσεων. Σκεφτείτε τις χτεσινές δηλώσεις του Υπουργού κυρίου Μωρατίνο από την απερχόμενη Προεδρία που από πολλές οπτικές ε, γωνίες πραγματικά θέλει να επιτύχει το αποτέλεσμα αυτό που είπε με σαφή ε, λόγια για τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Κούβα ότι στον τομέα αυτό προτιμότερε προτιμότερες είναι οι διμερείς συμφωνίες και όχι μια ξεκάθαρη ευρωπαϊκή θέση. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Κυρία, είπατε εκπρόσωπε, θα υπάρξει ένας σοβαρός κίνδυνος αν ενθαρρύνουμε αυτή την αμφισημία. Αν επιτρέψουμε να κρύβονται πίσω από την πολιτική συμφωνία η νιωστή διαπραγμάτευση μεταξύ κυβερνήσεων και όχι η, η υλοποίηση συγκεκριμένων μηχανισμών με αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Σβόβοντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι συγητές και ο κύριος Σεύκοβιτς και ιδιαίτερα η κάθε Άστον ε, κατάφεραν ένα πολύ καλό κείμενο να ετοιμάσουν. Η δική μου ομάδα ομόφωνα έλαβε γνώση και αύριο ε, με ομοφωνία και ομοψυχία θα υπερψηφίσουμε. Τώρα βέβαια μερικές κυβερνήσεις το βλέπουν ως ευκαιρία. Τώρα οι Γάλλοι έχουν άλλα προβλήματα με τις κόκκινες γραμμές, να τις αποσύρουν τις κόκκινες γραμμές. Πολλοί φοβούνται ε, στην κοινή γνώμη ότι θα αυξηθεί υπερβολικά η διπλωματία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα δεν πρόκειται για διπλασιασμό, αλλά για ενίσχυση των διπλωματικών υπηρεσιών. Ορισμένε κυβερνήσει θα υποχρεωθούν να αποσύρουν κάποιε διπλωματικέ υπηρεσίε όσο αναπτύσσεται η διπλωματική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλουμε. Ένα τέτοιο διπλωματικό σώμα. Και αυτό θέλουμε, κυρία Άστον, να δώσουμε ευκαιρία στη διπλωματική υπηρεσία μας και ελπίζω η Βελική Προεδρία να είναι η πρώτη που θα αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία. Και βέβαιως με τους υπουργού εξωτερικών και με τα ΙΠΕΞ, αλλά να έχουμε περισσότερη Ευρώπη στην εξωτερική πολιτική. Ο κύριος ε, λάμστορφ έχει το λόγο και εκπροσωπεί την ομάδα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Παραμονή της ψηφοφορίας θα πρέπει να κάνουμε ένα απολογισμό το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης δείχνει ε, ότι επιλέξατε μια καλή υποδομή, ένα προεδρείο και όχι μόνο ένα γενικό γραμματέα που θα ήταν παντοδύναμος και με πολιτική λογοδοσία και αυτό βοηθάει και στη συζήτηση και στην Ευρώπη και στις Βρυξέλλες για την εξωτερική διπλωματία αναβαθμίζει το επίπεδο και περιορίζει τη μονομέρεια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ενδιαφέρουν πάρα πολύ την ομάδα μου και χαιρόμαστε που έχω συμπεριληφθεί. Αλλά υπάρχουν και άλλα ε, πράγματα που μένουν να γίνουν. Δεν θελήσατε να έχετε μια μόνιμη πολιτική εκπροσώπηση. Βρήκατε κάποια λύση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά καμιά φορά διαφωνούμε. Αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι ο κόσμο ολόκληρο και θα πρέπει και στη Μαγιόρκα και στο Κίεβο, α πούμε, να ε, χρειάζεται να πάτε. Δεν μπορείτε να είστε πανταχού παρούσα. Και πώς θα το λύσετε αυτό. Είπατε, ε, κοιτάξατε τη ε, δήλωσή μου για την κεντρική διοίκηση. Μα έχουμε δύο δηλώσεις για την κεντρική διοίκηση. 48 ώρες μετά τη συμφωνία στη Μαδρίτη κάνατε δήλωση στο Κορεπέρ στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων και δεν ε, αφορά αυτό την απόφαση του Οκτωβρίου του 2009 μόνο, αλλά και το πρωτόκολλο 14 της ειδήξης Λισαβόνας που αντιφάσκει με αυτά που αποφασίστηκαν στη Μαδρίτη. Οπότε, δηλώσατε σήμερα και κάτι άλλο ακόμα στους εκπροσώπους ε, των λαών της Ευρώπης και ελπίζω αυτό να ισχύει και όχι αυτό που είπατε στις 23 Ιουνίου στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων. Δεν μπορείτε από τη μια να λέτε να έχουμε μια απαραίτητη δομή για την αντιμετώπιση των κρίσεων και από την άλλη να πηγαίνετε στο Κορεπέρ και να λέτε ότι εσείς θα είστε αρμόδιοι και μόνο. Ελπίζω να ισχύει αυτό που είπατε στο Κοινοβούλιο. Αυτό αντικαθιστά αυτό που είπατε στο Κορεπέρ. Και μην μου απαντήσετε ότι δήθεν δεν είναι αντιφατικέ μεταξύ του οι δηλώσει. Είναι σαφέστατο αυτό και τι θα πει, είτε η ενδεδειγμένη δομή, appropriate structure, το είπατε αυτό στα αγγλικά, θα φτιάξετε κάτι καινούριο, αλλιώς έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Χάουταλα για τους πράσινους. Θέλω να ευχαριστήσω, να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Ιδίω διότι λήφθηκαν απόλυτα υπόψη οι διαστάσει δικαιωμάτων του ανθρώπου ε, στην συμφωνία που επιτεύχθηκε και θέλω να παροτρύνω την ύπατη εκπρόσωπο να δράσει στηριζόμενη στη συμφωνία αυτή. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι γεννιέται μια στέρεη μονάδα, δυνατή μονάδα που θα προστατεύει τα δικαιώματα του ανθρώπου σε όλη τη διάσταση, σε όλες τις εξωτερικές ε, σχέσεις μας είναι σαφές ότι η διάσταση αυτή θα πρέπει να βρίσκεται ψηλά για να επηρεάζει την εξωτερική δραστηριότητα. Οι αντιπροσωπείε τη Ένωση προ τα έξω πρέπει να έχουν όλες υπεύθυνο δικαιωμάτων του ανθρώπου που θα ασχολείται με την επιτόπια υλοποίηση των θέσεών μα. Και επίση πρέπει να φροντίσουμε ούτω ώστε το Κοινοβούλιο, η υπηρεσία και οι ε, ύπατοι εκπρόσωπος να βρουν ένα νέο τρόπο συνεργασία που θα σέβεται το πνεύμα τη Λισαβόνα. Εμεί θέλουμε μια εξωτερική πολιτική πιο ισχυρή και πιο κοινοτική. Ο κύριος Τάνοκ έχει το λόγο. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης οδήγησε και προκάλεσε πολλές διαμάχες πρόσφατα. Ευτυχώς αυτή η διαδικασία έληξε και η κυρία Άστον έδειξε ότι, ότι έχει δεξιότητες για να ανταποκριθεί σε αυτό το έργο. Τώρα μιλάμε για ένα επικοδομητικό έργο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν και επικρίσεις. Ε, η ΕΕΔ αποτελεί μία αποδεκτή συμφωνία. Νομίζω όμως ότι μιλάμε για ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεν είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μία διακυβερνητική προσέγγιση και μία επιλογή ε, προσωπικού με βάση την αξιοκρατία. Και πιστεύω ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια πραγματική πολιτική και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα υπάρξει στελέχωση με το προσωπικό όπως προβλέπεται από τις συνθήκες. Τέλος, ελπίζω ότι οι εθνικοί βουλευτές θα συμμετέχουν ενεργά στη νέα αυτή διάρθρωση ελέγχου της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ιδιαίτερα ως προς τις στρατιωτικές αποστολές κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, που, γιατί τα κράτη είναι αυτά που χρηματοδοτούν τις πολιτικές άμυνας και ασφάλειας. Και αυτό αφορά ε, ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο που χρηματοδοτεί εμπολής αυτή την πολιτική μεταξύ άλλων κρατών. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος ε, Μάιερ από πλευράς Γκουε. Ευχαριστούμε κυρία Άστον, κύριε ε, Σεύκοβης. Αύριο δεν θα υπερψηφίσουμε την έκθεση αυτή για την ΕΙΕΒ, γιατί σε αυτή τη διαδικασία δυστυχώς υποκύψατε στις πιέσεις ορισμένων κρατών μελών. Και επίσης πιστεύουμε ότι τη στιγμή που αποφασίζεται αυτή η διάρθρωση δεν υπάρχει σωστή δομή ελέγχου αυτής της υπηρεσίας. Μιλάμε για ένα θεσμικό όργανο sui generis, σύμφωνα με το ε, οποίο θα υπάρχει έλεγχος από τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς το δημοσιονομικό έλεγχο. Εμείς είμαστε το μόνο θεσμικό όργανο που έχει εκλεγεί δημοκρατικά. Επίσης μας απασχολεί το γεγονός ότι οι στρατιωτικές αποστολές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της υπηρεσίας. Αυτό ε, αφορά το στρατιωτικό προσωπικό, την διαχείριση κρίσεων, χωρίς να ξεχνάμε και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Είναι μεγάλο λάθος που συνδέσατε τις, την υπηρεσία πληροφοριών με την ΕΙΕΔ, ιδιαίτερα σε σχέση με τα δημοσιονομικά μέσα και τον έλεγχό τους. Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να αποτελέσουν τμήμα αυτή τη υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων. Επίσης υπάρχει ένα στρατιωτικό σκέλος, ένα στρατιωτικός ε, προσανατολισμός που δεν δεχόμαστε. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια καθαρά πολιτική προσέγγιση χωρίς να είναι ουραγός του στρατιωτικού σκέλους. Θα έπρεπε δηλαδή να μας απασχολεί το θέμα της ανάπτυξης και της επίλυσης των σειράξεων. Γι' αυτό δεν θα υπερψηφίσουμε αυτή την έκθεση γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε προχωρήσει ως προς τον δημοσιονομικό έλεγχο, αλλά δυστυχώς τον τελευταίο λόγο δεν θα τον έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας μας οδηγεί και μας υποχρεώνει να καταψηφίσουμε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κάμπελ Μπάντερμαν, από την Ελευθερία και Δημοκρατία. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό που αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης που έχει σχέση με το διεθνές δίκαιο και τι σημαίνει κράτος. Σύμφωνα με την ε, συμφωνία του Μοντεβιντέο υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Κατερχήν μόνιμος πληθυσμός, ε, ορισμός της επικράτειας, κυβέρνηση και η δυνατότητα δημιουργίας διπλωματικών σχέσεων με άλλα κράτη το η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνιμο πληθυσμό τη συνθήκη της Λισαβόνας, άρα όλοι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, μία ε, συγκεκριμένη εδαφική ακαιρεότητα με συγκεκριμένα όρια, αν και το UKIP θεωρούσε ότι και το Συμβούλιο και η Επιτροπή αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας κυβέρνησης και διακυβέρνησης. Άρα μιλάμε για ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλα. Πιστεύω ότι ο ρόλος της Βαρόνης και με τη δημιουργία της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης πληρούνται όλα τα κριτήρια για να μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε με τη φωνή ενός κράτους. Μιλάμε για τα Ηνωμένα Έθνη της Ευρώπης. Υπάρχουν πολλοί υποστηριχτές και πιστεύω ότι αυτό επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου σε σχέση με την απειλή ως προς τα εθνικά κράτη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάρτογκ από τους μη γεγραμμένους. Σήμερα συζητούμε για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ε, το δικό κόμμα αντιτίθεται το κόμμα της ελευθερίας με κάθε μέσο κατά αυτές της υπηρεσίες διπλωματικής δράσης. Βγήκε από την αποτρόπαια συνθήκη της Λισαβόνας που με μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία και σωστά απέρριψε ολός της χώρας μου. Τελείως ε, αντιδημοκρατικό και με τρόπο ανεξέλεκτο κάνετε τώρα σχέδια για μια ευρωπαϊκή υπερδιπλωματία που θα... Ε, βγει προς τον κόσμο και όλη μεγαλύτερη εξουσία ε, σφετερίζεται από τα κράτη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυριαρχία δεν είναι στην Ένωση, είναι στα κράτη-μέλη. Τα σχεδιάκια της κυρίας Άστον θα επιβαρύνουν και την τσέπη του ε, φορολογούμενου. ο αεροπλάνο έχει για τον εαυτό τη και διάφορα εκατομμύρια αποζημίωση. Πού θα σταματήσει αυτή η ανοησία. Και έχει και ολόκληρη υπηρεσία που την πλαισιώνει και θα κάνετε ό,τι σας καπνίσει. Και ο πολίτης θα πληρώνει το αστρονομικό κόστος χωρίς να έχει λόγο. Αυτή είναι η δημοκρατία. Υπάρχει Ολλανδική πρεσβεία, προξενείο, ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στο εξωτερικό. Και ένας Ολλανδός που ταξιδεύει και βρεθεί σε δύσκολη θέση θα πρέπει να πάει στην πρεσβεία του. Μόνο αυτή ε, του δίνει μια υπηρεσία που θα είναι πραγματικά ε, λογική και σκόπιμη. Καταργήστε αυτή την υπηρεσία και αφήστε τη διπλωματία στα κράτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Λυπεί ομιλητέ. Που είναι στον κατάλογο. Ο κύριος Σαλαφράνκα Σάντσες Νέιδα για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε. Με την δήλωση τη ΥΠΑ τη εκπροσώπου και την ψηφοφορία αύριο ολοκληρώνεται η διαδικασία διαβούλευση. Άρα τώρα πρέπει να ευχαριστήσουμε του συναδέλφου για τη δουλειά που κατέστησαν κάτι τέτοιο δυνατό, ιδιαίτερα του ηγητέ του Κοινοβουλίου, να τηρήσουμε νομότυπα και να, το, και να υλοποιήσουμε τη συμφωνία για, χωρίς να ξεχνάμε ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δεν είναι αυτός σκοπός αλλά εργαλείο ούτως ώστε η Ένωση να μπορεί να διαθέτει μια εξωτερική πολιτική συνεκτική, ορατή και αποτελεσματική. Είμαι πεπισμένος ότι οι εγγυήσει ε, που έδωσε η κυρία Άστον στη δήλωσή της από την οπτική γωνία της πολιτικής ευθύνης είναι ικανοποιητικέ και συμπληρώνονται με τι αρμοδιότητε που αναφέρει η συνθήκη στο Κοινοβούλιο, τη διαδικασία ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή. Πρέπει να είστε βέβαιοι, κυρία Άστον, ότι το Κοινοβούλιο θα είναι ένα νόμιμ, νομιμόφρον εταίρο στην υλοποίηση της συμφωνία αυτής όπως ήδη δείξαμε στι συναντήσει που είχαμε με τους νέους επικεφαλεί των αντιπροσωπείων στην Όστιτον και την και το Αφγανιστάν. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε, κύριε Άστον, ότι η νέα υπηρεσία θα είναι πιο αποτελεσματική και καλύτερη από την υφιστάμενη. Εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, θέλω να σα ευχαρι... ευχηθώ καλή επιτυχία στην υλοποίηση τη της, ε, ε, ε υπηρεσία και να σα πω, όπω λέγει το Ευαγγέλιο, εκ των πραγμάτων κρυφίσεστε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σεβερίν, 1,5 λεπτό. Κυρίε και κύριοι, χρειαζόμαστε μια διενεργή εξωτερική πολιτική που θα καθορίζεται από τους στόχους μας και θα βασίζεται στις κοινέ μας αξίες. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζει το αδιέρετο της ασφάλειας σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο ως πηγή αλληλεγγύης και συμφερόντων εντός και εκτός Ένωσης. Μια τέτοια πολιτική που έχει στόχο την αύξηση της ικανότητας της Ένωσης να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες της και να βελτιώνει την δυνατότητα της να διαμορφώνει το παγκόσμιο περιβάλλον και όχι μόνο να αντιδράσει σε αλλαγές, απαιτεί σωστή θεσμική πλαισίωση και αποτελεσματική υπηρεσία εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Μην ξεχνάτε ότι ε, η υπηρεσία αυτή δεν είναι όργανο απόφασης αλλά μια, ένα κοινοτικό εργαλείο που εφαρμόζει την κοινοτική πολιτική στην εξωτερική δράση και να, να διευκολύνει νωρίτερα την λήψη σχετικών αποφάσεων υπό την εξουσία της Αντιπροέδρου και σε συντονισμό με, με τους άλλους παράγοντες οι βασικές ανησυχίες του Κοινοβουλίου ήταν σαφείς. Να υπάρχει πολιτική παρακολούθηση, λογοδοσία και από την δημοσιονομική διάσταση. Αυτό απαιτεί διαφάνεια στη λειτουργία της υπηρεσίας και σαφήνεια μέσω της παρουσίασης ενός ενοποιημένου προπολογισμού της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να ελέγξει το Κοινοβούλιο κατά πόσο τα μέσα ε, αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές και πόσο αποτελεσματικές είναι οι πολιτικές αυτές. Δεν χρειάζεται να αναφέρω περισσότερο για τα ζητήματα αυτά. Παρέχεται, καλύπτονται οι ανάγκες μας ε, και παρέχεται δυνατότητα αναθεώρησης που θα προβλέπει την ε, πύληση των ε, προβλημάτων που ανακύπτουν ευνίδια. Διακόπτεται ο, ο ο μιλητής από τον πρόεδρο. Ο επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Νταφ. Πρόεδρε, από ό,τι φαίνεται υπάρχει ευρεία συμφωνία για τα μέσα, τις διεργασίες και το προσωπικό. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα επιχείρημα για διαμόρφωση πολιτικών που θα είναι επαρκώς θαραλέο για να μπορούμε να συγκρίνουμε, να αντιπαραθέτουμε και να αμφισβητούμε την εθνική εξωτερική πολιτική. Εάν αποτύχουμε στην παρουσίαση των επιχειρημάτων αυτών δεν θα αναδυθεί μια πραγματικά κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Πιστεύω λοιπόν ότι η κυρία Άστον θα πρέπει να, διαφ... να θέσει και να απαντήσει σε μια σειρά σκληρών ερωτημάτων. Για παράδειγμα, γιατί ακόμα πέντε κράτη αρνούνται να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία του κοσμοπεδίου. Γιατί η Ελλάς επιτρέπεται να παρεμποδίζει την εμφάνιση της Μακεδονίας ως κράτους. Γιατί υπάρχει ακόμα ψυχρός πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου. Ελπίζω, εάν θέσει αυτά τα σκληρά ερωτήματα, να παράσχει και κάποιες δημιουργικές και θαραλέες προτάσεις λύσης. Για παράδειγμα, την πρόταση να ξεκινήσει μια κοινή αποστολή κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας για την καταπολέμηση του, του οργανωμένου εγκλήματος. Κάτι τέτοιο είναι η μορφή πολιτικής που επιζητούμε αυτή τη στιγμή από την κάθε άστον και τις υπηρεσίες της που θα είναι υπηρεσίες άριστης διπλωματίας. Καλή τύχη και ευχαριστούμε για τις μέχρι τώρα επιτυχίες σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σαρτζεντίνη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Οι εκπρόσωποι των Πρασίνων μίλησαν για το στοιχείο εκπροσώπησης των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Εξωτερική Δράση γενικά. Εγώ θα ήθελα να τονίσω την αναπτυξιακή συνεργασία ε, ως ευρωπαϊκό σχέδιο. Ο κύριος Κάσμαρεκ, αρμόδιος συζητητής της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας, δεν θα πρέπει να είναι ένα κίνητρο μόνο που να χρυσώνει το χάπι για να βρίσκει το δίκιο της η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παγκόσμια. Θα πρέπει να υπάρχει μια πραγματική δομή στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και αναπτυξιακή Όμω, συνεργασία να είναι ευθύνη του Επιτρόπου Πίμπαξ, να παραμένει εκεί και να φροντίζει να είναι συνεκτική η πολιτική και εμεί, οι πράσινοι θα τον βοηθήσουμε στην προσπάθεια αυτή να φροντίσει η εξωτερική μας πολιτική κυρίως να στρέφεται στην καταπολέμηση της φτώχεια. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you, madam. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φόξ. Η κυρία Φόξ, με συγχωρείτε, that είχα αντιταχθεί στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θεωρώ ότι η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να αποτελέσει προνόμιο, αποκλειστικό προνόμιο των κρατών μελών αλλά ως πραγματιστής θα πρέπει να αντιμετωπίσω την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι και όχι όπως θα ήθελα να είναι. Γι' αυτό καλωσορίζω την εξαιρετική συνεργασία των εισηγητών σε συνεργασία με την Βαρόνη Άστον. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία όπου θα υπάρχει και δημοσιονομικός έλεγχος της υπηρεσίας. Επειδή ζούμε σε εποχή λιτότητας δεν θα πρέπει να γίνουν υπερβολικές δαπάνες, δηλαδή μέσα στα πλαίσια της κατάρτισης διπλωμάτων. Όπω όπως συμβαίνει συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βαρόνι Άστον μας είπε ότι θα είναι η υπηρεσία δημοσιονομικά ουδέτερη. Δεν νομίζω ότι θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο, αλλά αν θέλουμε να τιμήσουμε τους φορολογούμενους, θα πρέπει να τη ζητήσουμε να τηρήσει αυτή την υπόσχεση. Ευχαριστούμε. Πέλντερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο λόγους για τους οποίους θα καταψηφίσω την έκθεση Block και Χόφστατ. Είναι νοσηρή αυτή η δίψα τους για ε, εξουσία. Αρκεί να συμμετέχει το, κοινοβούλιο και όλα εντάξει. Και η κυρία Άστον, γιατί χρειάζεται τέτοια υπηρεσία. Το δεύτερο αφορά το πού θα μπει αυτή η υπηρεσία θεσμικά. Τους τελευταίους μήνες φάνηκε ότι η διπλή ιδιότητα είναι ένα πείραμα θεσμικό και δεν είναι μεγάλη επιτυχία. Και έχουμε και μερικές τώρα χιλιάδες διπλωμάτες που θα έχουν διπλή ιδιότητα. Οποίο θέαμα. Και που αυτή είναι μια φαιά ζώνη. Ε, είναι και δεν είναι στην Επιτροπή, δεν λειτουργούν τα πράγματα καλά, δεν πάει καλά αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φιλίπ Κλάς. Για ένα, ε, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα λόγου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ο έλεγχος γίνεται κυρίως από τον προϋπολογισμό και κατά τα άλλα είπα ότι εκπρόσωπος θα πρέπει να λογοδοτεί στο κοινοβούλιο. Μα αυτό είναι το φυσιολογικότερο πράγμα του κόσμου. Σε μια δημοκρατική πραγματικότητα, ή ε, αυτό που πρέπει να είναι δημοκρατικό σύστημα. Τώρα έχουν δημιουργηθεί και προσδοκίες για τους πολίτες και ελπίδες ότι θα έχουμε λέει μια ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία. Αλλά εάν στα κράτη-μέλη τα ίδια δεν υπάρχει κοινό όραμα, τότε είναι κενό γράμμα η διπλωματική υπηρεσία. Τι να την κάνουμε θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στο μήνυμα, αλλά δεν είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Είδα και στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου ένα άρθρο με τίτλο «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρνει πιο κοντά στους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Διπλωματική Υπηρεσία». Πώς ακριβώς θα γίνει, δυστυχώς δεν το εξηγεί αυτό το άρθρο. Είναι μια κενή προπαγάνδα, γιατί όλο και περισσότεροι πολίτες μας γυρίζουν την πλάτη. Ευχαριστώ. Κύριο κύριος Γιάτσο Βόλσκι. Uh, Ευχαριστώ. Κυρία Ήπατη, εκπρόσωπε, πολλές φορές ίσως θα ήταν σκόπιμο να μιλάμε για τον για τίτλο του Υπουργού Εξωτερικών. Η ΕΙΕΔ έφτασε πια στο προσκήνιο. Ήταν κάτι που αναμέναμε εδώ και πολύ καιρό και θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, να μιλάμε με μία φωνή σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αλλά επίσης θα πρέπει να κινηθούμε πέρα από τις λεπτομέρειες και τις τεχνικές διευθετήσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, χωρίς να υπάρχει δημοκρατική ε, νομιμότητα, η η υπηρεσία εξωτερικών, εξωτερικής δράσης δεν θα είναι αποτελεσματική και σωστή. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ε, σοβαρός έλεγχος των επιλογών εξωτερικής πολιτικής. Θα πρέπει να έχουμε μια δυνατή υπηρεσία και να εκπροσωπεί και τα 27 κράτη-μέλη. Μεγάλα, μικρά, παλαιά και νέα από το βορρά προς τον νότο, από ανατολάς προς δυσμάς να λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή, ε, κοινή μια σωστή αναγνώριση με μια σωστή γεωγραφική κατανομή. Πιστεύω με την απόφαση του Συμβουλίου θα γίνει πιο κοινοτική η υπηρεσία, θα μας εκπροσωπεί γεωγραφικά και εθνικά. Και επίσης με το δημοσιονομικό κανονισμό θα υπάρξει νέα και σωστή κατανομή εξουσιών για να βελτιώσουμε την ε, ΕΕΔ. Ο κύριος Βιγγένιν για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Λέδι Άστον, συνάδελφοι, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη σύσταση αυτής της υπηρεσίας η οποία ε, δημιουργούσε πολλές αμφιβολίες ως προς τη σύσταση της έξι μήνες πριν. Δεν ξέραμε κατά πόσο η Λέδη Άστον θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες προκλήσεις και ευθύνες. Νομίζω ότι αυτές οι αμφιβολίες ήταν βάσιμες και η Λέδη Άστον κατάφερε να ε, φτάσει στη σύσταση αυτής της ε, υπηρεσίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάστηκε ευθύς εξ αρχής για τη σύσταση αυτής της υπηρεσίας και θα προβάλλουμε και τροπολογίες ως προς το δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. Η γεωγραφική κατανομή είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας γιατί υπάρχουν ορισμένα κράτη που δεν εκπροσωπούνται σωστά σε αυτή την ε, ιεράρχηση που γίνεται. Εγώ εκπροσωπώ μία από αυτές τις χώρες και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τη, την αντίρρησή μου ως προς, τις αντιρρήσεις μου ως προς αυτό το σκέλος. Επίσης, τα νέα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν ένα έργο κατάρτισης των διπλωματών τους, έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικά και πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει καμία κατάχρηση εξουσίας από την Ε.Ε. για να επιλύσει καθαρά ε, εσωτερικά εθνικά ζητήματα. κύριος Γκέρενς, λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Έλμαρ Μπρόκ και τον Γκίφερ Χόφστατ, διότι κατόρθωσαν να παρουσιάσουν και να κερδίσουν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής με ένα πραγματικό πολιτικό, με μια πραγματικά πολιτική προσέγγιση. Επίσης να ευχαριστήσω τις προσπάθειές τους για τη διαφύλαξη μιας ενιαίας προσέγγισης στην πολιτική ανάπτυξη και συνεργασία. Η θέση του Επιτρόπου Πίμπαλξ για την ε, για τη συνεργασία και της κυρίας Δημήτρεβα για την ανθρωπιστική δράση είναι καθοριστικές για να υπάρχουν φυσικές δραστηριότητες της Ένωσης του τομείς. Βεβαίως να επιτύχουμε συνεργεία μέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Ε, είναι αναγκαίο κάτι τέτοιο, όπως είναι εξαιρετικά επιτακτικό να μιλάμε με μία φωνή. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτός που μιλά εξ ονόματος της Ένωσης να μην ε, διαψεύδεται από αυτά που λέει ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης. Δεν ξέρω αν όλοι έχουν καταλάβει το μήνυμα σήμερα. Για να το καταλάβουν χρειάζεται μια πραγματικά ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Μεγάλη πρόκληση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε απόψει για τα μεγάλα ζητήματα. Μία άποψη για τα μεγάλα ζητήματα του κόσμου, για την Τουρκία, για το Ιράκ, για όλα τα ζητήματα για τα οποία ε, θα πετύχετε κάτι τέτοιο κύριε είπατε εκπρόσωπο θα έχετε τις επιδοκιμασίες της ε, ε, συνέλευσής μας. Ο κύριος Πιωτόφσκι, ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής δράση είναι ο καρπός της συνθήκης της Λισαβόνας. Σε πολλά κράτη-μέλη, ωστόσο, δεν έγινε δημοψήφισμα και οι Ευρωπαίοι πολίτε κατά συνέπεια δεν μπόρεσαν να πούνε αν συμφωνούν ή όχι με την υπηρεσία αυτή. Εμά μα ανησυχεί πολύ το γεγονός αυτό, διότι έχουμε την εντύπωση ότι στην πράξη είναι η, γίνεται μια διαμάχη μεταξύ χωρών, κάποιων χωρών για να έχουν τι καλύτερε θέσει στην αυτή υπηρεσία. Γι' αυτό ζητούμε να υπάρχει και γεωγραφική ε, εξισορρόπηση. Επίση, δεν θεωρούμε ότι η υπηρεσία αυτή πρέπει να απομονωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια. Πιστεύω ότι πρέπει τα κράτη-μέλη να μετάσχουν ουσιαστικά στην άσκηση ελέγχου στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και να αποκτήσει η υπηρεσία αυτή ουσιαστική νομιμοποίηση. Κάτι που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, διότι αποκλείεται από τη διαδικασία το εθνικό, τα, αποκλείονται τα εθνικά κοινοβούλια. Ε, επίσης, μέσα σε αυτά τα πλαίσια κρίσης που ζούμε χρειάζεται να επενδύσουμε σε μια τέτοια υπηρεσία. Ο κύριος Ντανζόν, 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Άστον, θα ήθελα να σας εκφράσω την υποστήριξή μας χωρίς καμία αμφιβολία ε, ως προς αυτό το συμβιβασμό Μπροκ, Φερχόφστατ, Πρόκειται για μια κοινή πολιτική σε θέματα ασφάλειας, άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και είναι η πολιτική που βλέπουμε σήμερα από τη Σομαλία μέχρι τη Γεωργία από... και μέχρι τη Γάζα και είναι κάτι το οποίο επιθυμούσαν οι πολίτες μας. Δεχόμαστε αυτό τον διαθεσμικό συμβιβασμό με τις αυξημένες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτός ο φορέας είναι χρήσιμος για να έχουμε μια συνεκτική και αξιόπιστη καθώς και αποδοτική πολιτική εξωτερικών σχέσεων. Επειδή συμμετέχω στην ε, Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας και ως Γάλλος θα ήθελα να δω ότι προσδίδω μεγάλη σημασία στις ευθύνες σας ως προς τη διαχείριση κρίσεων, ενισχύοντας ε, την προστιθέμενη αυτή αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την σύμπραξη πολιτικού και στρατιωτικού σκέλους. Εσείς θα πρέπει να εγγυηθείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει και θα αυξήσει τις δυνατότητές της έτσι ώστε να διασκορπιστούν οι αμφιβολίες σε σχέση με την στρατιωτικοποίηση της υπηρεσίας και ε, με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου για, την για τον έλεγχο της ε, νομιμότητας όλων των πράξεων και δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χάουιτ, για ένα λεπτό. Θα ήθελα να συγχαρώ την Κάθη Άστον και τους συναδέλφους, διότι φτάσαμε σε ένα συμβιβασμό για το όραμά μας για αυτή την ολοκληρωμένη Ευρώπη που θα αφορά όλες τις δραστηριότητες και προνόμια και αρνούμενη τα στοιχεία που είναι υπέρ γραφειοκρατικών αυτοκρατοριών. Εκείνοι που ανησυχούν για την εθνική εκπροσώπηση θα πρέπει να υποστηρίξουν την Βαρόνη έτσι ώστε να γίνουν διορισμοί με βάση την αξιοκρατία. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι, το, αυτός είναι ο απότερος στόχος για να κοιτάμε το μέλλον και όχι το παρελθόν και να μην έχουμε νεοαπικιακή προσέγγιση στο όλο θέμα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφασιστεί ε, αυτό το σχέδιο και να ενταχθεί στη, στο δημοσιονομικό μας κανονισμό, διότι σε λίγο θα κλείσουμε και τον ένα χρόνο διορισμού της ΥΠΑ της εκπροσώπου. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το προωθήσουμε αυτό, Βαν Πολύ αντιταχθήκαμε στην ιδέα μιας υπηρεσίας εξωτερικής δράσης γιατί είναι μία ε, ολέθρια συνέπεια της συνθήκης της Λισαβόνας και της ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που δεν επιθυμούν ε, πολύ από εμάς. Ε, εγώ όπως και ο Βρετανός ΥΠΕΞ αναγνωρίζω την ύπαρξη της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ως γεγονός. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα θέλαμε η ύπατη εκπρόσωπος να μας δώσει εγγυήσει ως προς την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, ότι δεν θα δημιουργήσει σε επιπρόσθετο κόστος, δεν θα παρέμβει ή δεν θα μειώσει το ρόλο των εθνικών διπλωματικών ε, αντιπροσωπιών, ιδιαίτερα του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης ότι δεν θα είναι ένας επιπρόσθετος γραφειοκρατικός οργανισμός και θα την χάνει της επίβλεψης των Εθνικών και του παρόντος Κοινοβουλίου. Επ' αυτού θα ήθελα να πω ότι επειδή φέρει ευθύνη και για την πολιτική άμυνας και ασφάλειας και ε, επειδή η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση έχει διαλυθεί, πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες και στον τομέα της άμυνας της ασφάλειας. Και επειδή οι στρατιωτικές δυνάμεις υπόκεινται στο εθνικό... Ε, ε Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Κάσπαρη για 1,5 λεπτό. 1,5 λεπτό λέει ο κύριος Κάσπαρη. Ελπίζω να ακούσετε το τέλος της παρέμβασής μου, λέει ο κ. Βανόντεν. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο κ. Κασπαρή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση είναι ακόμα ένα βήμα προ μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Θεωρώ την υπηρεσία αυτή τεράστια ευκαιρία. Και σα εύχομαι, αξιότιμη κυρία Άστον, ε, καλό κουράγιο και δύναμη ε, στο έργο σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Έλμα Μπρόκ και όσου αγωνίστηκαν μαζί του το τελευταίο διάστημα, του τελευταίου μήνε, οι διαπραγματεύσει κατάφεραν να πετύχουν πολλά, όχι μόνο για το Κοινοβούλιο, αλλά για του πολίτε κυρίω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υποδειγματική. Θα ήθελα να μιλήσω για το εξωτερικό εμπόριο. Σε αντίθεση με την ΚΕΠΑ, Υπάρχει ήδη κοινή εξωτερική πολιτική εμπορίου εδώ και δεκαετίε, με πολλέ θετικέ εμπειρίε στο εξωτερικό εμπόριο. Και αυτά μπορούν, νομίζω, να μεταφερθούν και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Θα επιθυμούσα όμω ρητά Εκεί και στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης στο μέλλον να μην επισκιάσει ή να μην μπλοκάρει άλλες πολιτικές όπως είναι η εμπορική πολιτική. Εδώ θα χρειαστεί να λυθούν κάποια πράγματα στις λεπτομέρειες. Θα ήθελα να σας παραπέψω στην γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου του συναδέλφου Σαχραντή και από την ομάδα μου ο κύριος Αλέσκη το έχει ε, υποστηρίξει πολύ και θα Χαιρόμουν πάρα πολύ αν υπαλληλή σα βαρώνει τα λάμβαναν αυτά υπόψη το επόμενο διάστημα στην εργασία τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπέρμαν έχει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Τες Μπέρμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε λίγους μήνες άλλαξαν πολλά για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Τον Ιανουάριο στην Ακρόαση για τους νέους Ευρωπαίους Επιτρόπους εγώ με την ομάδα μου εξέφρασα κριτική ότι ο Επίτροπος για την Αναπτυξιακή Βοήθεια κανονικά γίνεται μάνατζερ για ένα τμήμα μόνο ε, του τομέα του χωρίς οι ίδιες ευθύνες. Η αναπτυξιακή βοήθεια υπόκειται σε κριτήρια ε, εξωτερικής πολιτικής και εμπορικά με κοινικό τρόπο όπως έκανε δικτάτορες εδώ και δεκαετίες εις βάρος του πληθυσμού. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Βέβαια είναι φυσικό να υπάγεται και αναπτυξιακή πολιτική στην εξωτερική πολιτική με εποπτεία της Ελέδης Άστον αλλά με συγκεκριμένο στόχο, συγκεκριμένη χρηματοδότηση και ξεχωριστή πολιτική. Μόνο έτσι μπορεί να παίξει το ρόλο που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της φτώχεια και τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η δική μας πολιτική ομάδα θα φροντίσει αυτό να προωθεί και μπορεί να γίνει με την παρούσα υπηρεσία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πορέμπα, ένα λεπτό. Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο συνέβαλε με επικοδομητικό τρόπο στην επίτευξη μιας συμφωνίας. Νομίζω ότι το πετύχαμε στον τομέα που συζητούμε σήμερα. Αλλά πρέπει να υπενθυμίσω ότι τα κριτήρια που πρέπει να καθοδηγούν τη ε, στάση μας στην υπηρεσία είναι επαγγελματισμός, αλλά ταυτόχρονα και γεωγραφικά κριτήρια. Να περιλαμβάνουμε διπλωμάτες από τα νέα κράτη-μέλη, που μπορεί να μην έχουν μεγάλη εμπειρία στα θεσμικά όργανα της Ένωσης όσο και τα παλιά, αλλά που έχουν και καλή προαίρεση και ανάγκη να παρίστανται στην υπηρεσία αυτή. Αυτό σας υπενθυμίζω σήμερα κυρία είπατε εκπρόσωπε. Πρέπει να ανοίξετε τις πόρτες της υπηρεσίας σε Σλοβάκους, Ούγκρους, Πολωνούς για να ενισχύσετε την νομιμοποίηση της υπηρεσίας αυτής. Χαίρο λοιπόν για την δημιουργία της υπηρεσίας αυτής. Πρέπει να δείξετε ωστόσο αποφασιστικότητα και σταθερότητα. Διακόπτεται ο μιλητής. Η κυρία Γκρέσλε, 1,5 λεπτό. Frau Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, συγχαρητήρια ε, για την ίδρυση της 28ης διπλωματικής υπηρεσίας. Βαφτίζουμε ένα νέο σώμα χωρίς να ξέρουμε ε, το επιτελείο, το κόστος, της υπηρεσίας που θα παρέχει. Τι σημαίνει, πόσο είναι το γρανόγραμμα, γιατί έχουμε και συμβασιούχους και ε, ε χώριους Έχουμε μια αρχιτεκτονική που έχει μεγάλες αδυναμίες και που ελέγχεται ε, δυσκολότερα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή υπηρεσία. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι σας πιστεύω ειλικρινά ότι ε, θέλετε να αναγνωρίσετε το δικαίωμά μας για τον προπολογισμό και την εξουσία μας για τη χορήγηση της απαλλαγής, αλλά να πείσετε το Συμβούλιο ε, ότι χρειαζόμαστε τη δήλωση αξιοπιστίας του Ευρωπαίου Πρέσβη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το δημοσιονομικό κανονισμό. Επίσης θα σας παρακαλούσα το, ε, τις διοικητικές δαπάνες του οικοδομήματος αυτού να τις μειώσετε χρησιμοποιώντας ε, τις δομές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν το κάνετε παρκώς οφείλουμε στους πολίτες να επιλέγουμε τις πιο φτηνές δομές και συλλοποίηση των πολιτικών μας να έχουμε οικονομίες. Δημοσιοποιήστε παρακαλώ το κόστος. και να σταματήσουν οι αψημαχίε και οι διαπληκτισμοί μεταξύ των ίδιων των υπαλλήλων σας για να έχει και αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βόλφκαν Κράισερ Ντόφλερ για ένα λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κοινή εξωτερική πολιτική στην Ένωση χρειαζόμαστε επιγόντως. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι πολλά τα εμπόδια. Για τον κανονισμό του προσωπικού ε, και το δημοσιονομικό κανονισμό θα πρέπει να γίνουν δεκτά αυτά που ζητάμε. Και ορισμένοι κυβερνώντες και υπουργοί εξωτερικών θα πρέπει να βάλουν κάποια στιγμή στην άκρη τα δικά τους συμφέροντα, να υποτάξουν στο κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον τα εθνικά. Καλωσορίζω το γεγονός ότι θα έχουμε μεγαλύτερο ρόλο για την αυτοξιακή πολιτική, για την πολιτική γειτονία που παραμένει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει από ποιο κράτο μέλο προέρχονται οι υπάλληλοι τη υπηρεσία εξωτερική δράση. Η αξιοκρατία είναι το κριτήριο. Όχι αν είναι ο άλλο Πολωνό, Γάλλο ή Γερμανό και μιλάει τη μητρική του γλώσσα θα πρέπει ε, ε, οι πολίτες αυτοί, οι διπλωμάτες αυτοί να αισθάνονται υπόλογοι στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία και όχι στα Υπουργεία Εξωτερικών τους. Αυτό περιμένουν οι πολίτες από εμά. Συνεργασία, ε, μπορείτε να υπολογίζετε και καλή τύχη. Επικοδομητική πάντα, αλλά και με κριτικό πνεύμα. Κύριο Ξύπ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία είπατε εκπρόσωπε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την έκθεση που οδήγησε σε αυτό το συμβιβασμό έτσι ώστε μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης που ελπίζω να εγκριθεί αύριο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τη δημιουργία αυτής της υπηρεσίας ε, υπάρχουν πολλές ελπίδες, υπάρχουν και πολλές προτεραιότητες. Θα πρέπει να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αναπτυξιακή πολιτική. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της εγγύησης της γεωγραφικής εκπροσώπησης της σωστής γεωγραφικής εκπροσώπησης. Έτσι όλα τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα τα νέα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να κατανοήσουν ότι αυτή η υπηρεσία δημιουργήθηκε για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω αυτή η απόφαση να τηρηθεί και από το Συμβούλιο. Ο κύριος Γκάλερ για δύο λεπτά. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Γενικά συμφωνώ με το συμβιβασμό κοινοτική μέθοδος διατηρείται, αποκρούστηκε η απόπειρα του Συμβουλίου να το παρακάμψει αυτό και παραμένει κοινοβουλευτικός έλεγχος. Παραμένουν βέβαια κάποιες ε, λεπτομέρειες να λυθούν ε, στο δημοσιονομικό κανονισμό. Ε, θέλω να ζητήσω το εξή από εσά προσωπικά. Και στην εξωτερική πολιτική θα πρέπει να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που έχετε. Έχω την εντύπωση ότι δεν έγινε αυτό στο παρελθόν όσο θα μπορούσε να γίνει. Η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βελτιωθεί παντού. Και στην εξωτερική πολιτική θα πρέπει να κατεβαίνουμε καμιά φορά και από το θάλαμο διακυβέρνησης στους σκάφους ας πούμε στις μηχανές να φεύγουμε από την Επιτροπή Εξωτερικών και να βλέπουμε τι γίνεται στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, εκεί στο μηχανοστάσιο. Ευχαριστώ. κυρία Σουζάννα Ρόιτοβα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την συμμετοχή των 27 κρατών μελών. Ο κύρι, οι κύριοι Φερχόστατ και Μπρόκ ε, προετοίμασαν περισσότερα από 70 τροπολογίες έτσι ώστε να προωθηθούν τα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα και όχι τα εθνικά. Έχει μεγάλη σημασία και το πρόγραμμα χρηματοδότησης Διακόπτη ο μιλητής, ομιλήτρια. Νομίζω ότι τα χρήματα θα πρέπει να καταβληθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και για το 1 τρίτον των υπαλλήλων που θα διοριστούν από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να συμφωνήσω με την ύπατη εκπρόσωπο ότι οι διπλωμάτες θα πρέπει να έρθουν πρώτοι, αλλά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει μια σωστή γεωγραφική εκπροσώπηση διπλωματών και μόνιμου προσωπικού. Εάν θέλουμε όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν αναλογικά στην ΕΙΕΒ, θα πρέπει να κάνω μία έκκληση προς την Κομισιόν οι υπηρεσίες να μην υπηρετούν τα μεγάλα κράτη-μέλη. Πάτε πολύ γρήγορα. Τι? Αν μιλάτε πολύ γρήγορα, δεν σα προλαβαίνουν διερμηνείς. διερμηνεί. Μιλήσετε ένα και 20 και είχατε 1,5 λεπτό. Μπορούσατε να είχατε μιλήσει πιο αργά για να μεταφραστείτε και καλύτερα. Ο κύριο Ζαλεύσκη, για ένα λεπτό. Πάνι Άστον, ε, το ε, Κυρία ε, Άστον, αύριο θα πρέπει να αποφανθούμε επί ενός σημαντικού έγγραφου που θέτει τις βάσεις για τη λειτουργία της ΕΙΕΒ. Πρόκειται για μια πραγματική ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία και ε, χάρη της συνθήκης της Λισαβόνας προβλέπεται αυτή η δυνατότητα. Είχαμε εκφράσει πολλές ανησυχίες βεβαίως εξ αρχής, γιατί θέλαμε να ξέρουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες της κυρίας Άστον έναντι ορισμένων μεγάλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναρωτηθήκαμε κατά πόσο θα είχατε αρκετά περιθώρια ελιγμών, διότι ορισμένα κράτη-μέλη είναι πολύ επιφυλακτικά ως προς το να εγκαταλείψουν ορισμένες εθνικές αρμοδιότητες. Θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή γεωγραφική κατανομή και κάνω μια έκκληση προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Όμεν για ένα λεπτό. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όχι μόνο τον συνάδελφο Αλμαρ Μπρόκ, αλλά και τον συνάδελφο Φερχόφστατ που αγωνίστηκαν και οι δύο για να έχει Ευρώπη ενιαία φωνή στον κόσμο και δυνατή. Θέλω πω το συνάδελφό μου από το κόμμα της Ελευθερίας, το ΠΒΒ της Ολλανδίας, ότι στην συντακτική συνέλευση και το Ολλανδικό κράτος αγωνίστηκε για ενιαία ε, εξωτερική δράση και υπηρεσία. Τι έχουμε πετύχει. 75 αλλαγές από την αρχική πρόταση του Συμβουλίου. Δεν είναι διακυβερνητικό όργανο, αλλά είναι κοινοτική μέθοδος. Πλήρω συμμετέχει το Κοινοβούλιο και για τον προπολογισμό και για τη στρατηγική και ε, για τους πρέσβεις. 60% ε, των ε, διπλωματών είναι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα έρχεται η δοκιμή. Εσείς κυρία Άστον θα πρέπει να φροντίσετε με την υπηρεσία σας αυτή να είναι ενιαία η φωνή της Ευρώπης στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσε ο χρόνος σας. Καλά καλά λέει η κυρία Όμεν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κάτσε διάει. Κύριε Κολάνσκα Μπαμπίνσκα για ένα λεπτό. Κυρία Άστον, πιστεύω ότι η υπηρεσία εξωτερικής είναι ένα βήμα μπρο για την ενίσχυση της εικόνας της Ευρώπης και πιστεύω ότι θα συμβάλλει στην επίτευξη των σημαντικών στόχων της Ένωσης και των κρατών μελών και στον τομέα της ενέργειας. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει εξειδίκευση στους διάφορους τομείς. Δεν πρέπει η υπηρεσία αυτή να είναι μόνο μια ασαφής διπλωματική υπηρεσία πιστεύω ότι θα έπρεπε να προσλάβει ειδικού που γνωρίζουν καλά πολιτική ενέργειας, πολιτική ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε μια ευέλικτη λοιπόν δομή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο κριτήρια γεωγραφικής εκπροσώπησης, αλλά να μπορούμε να προσλάβουμε ανθρώπους που δεν δουλεύουν στο δημόσιο ανάγκη. Τα κριτήρια αυτά αναφέρθηκαν και από μη κυβερνητικούς οργανισμού. Είναι σημαντικό για να πετύχουμε τους στόχους μας να τηρήσουμε τις ε, ε, προϋποθέσεις αυτές. Ο κύριος Πάσκου για ένα λεπτό. Thank you, Mr. President. The creation of... Ευχαριστώ. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης είναι ένα πολύ καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης θα αλλάξει το εν γέννη σχήμα μας ε, ως προς την χαμηλότερη χρήση της γραφειοκρατίας. Μιλάμε για μια κοινή εξωτερική πολιτική. Θα ήθελα να μιλήσω για το χάσμα μεταξύ των προσπαθειών μας ώστε να χορηγήσουμε μια σωστή νομική ε, βάση στην υπηρεσία και την πραγματικότητα της στελέχωσης γιατί μιλάμε για γεωγραφική κατανομή και ήδη γίνονται συνεντεύξεις για προσλήψεις και από ε, τα νεα κρατημένη φαίνεται ότι δεν υπάρχει ε, μεγάλη ελπίδα για αυτούς, για τους υποψηφίους, από τα νέα δηλαδή. Γι' αυτό με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι αρχές αυτές θα πρέπει να τηρηθούν όμως και όσο το νωρίτερο τόσο το καλύτερο. Κύριος Βάιγκλ, ένα λεπτό. Κυρία Άστον, χτες το Κοινοβούλιο άκουσε έναν κύριο που δεν είναι διπλωμάτης, που δεν είναι πολιτικός, τον κύριο Τζον Γκίντ, εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Γάζα. Μας είπε πολλά πράγματα στην, για την Γάζα και μας είπε και για τον κύριο Μπλερ, δεν, ξέρει, ξέρουμε τι κάνουμε εκεί. Μας είπε ότι υπάρχουν υπουργοί εξωτερικών που δεν θέλουν να επισκεφθούν τη Γάζα. Θέλω να πω το εξή. Σα συγχαίρω για την δημιουργία της υπηρεσία αυτής και για τις προσπάθειες που καταβάλλετε εσείς και οι συναδελφοί σας για να γίνει η υπηρεσία αυτή αποτελεσματική. Θα είναι ωστόσο αποτελεσματική αν είναι δημιουργική και τούτο εξαρτάται από την ε, πνευματική επίδοση των υπαλλήλων σας. Θα ήθελα και εύχομαι να έχετε μια ομάδα ισχυρών δημιουργικών ανθρώπων. Ευχαριστώ Πρόεδρε θα ήθελα ε, να πω ότι είναι καλή η είδηση αυτή στην Ευρώπη όταν έχουμε οικονομική και καμιά φορά πολιτική κρίση, λέει ο κύριος Λόπες Ιστούρης. Έχουμε ε, κάνει καλά βήματα προ τη σωστή κατεύθυνση για την υπηρεσία εξωτερική δράση. Θέλω να ευχηθώ όχι μόνο στην ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο αλλά και σε όλου του άλλου πρωταγωνιστέ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον καλό μα φίλο Έλμαρ Μπρόκ που διευκόλυναν τι συμφωνίε για να φτάσουμε σε εκεί. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε κυρία Άστον ότι αυτό που θα πρέπει να υπερασπιστούμε κυρίω είναι τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα λέω και δεν είναι συμβούλη, απλώ ένα σχόλιο. Με τα, όσα είπε ο Χωσέ Ιγνάσιος Αλαφράγκα, καλός μου φίλος και ε, αυτό που χρειάζεται είναι αποτελεσματικότητα και εγώ θα πρόσθετα και ε, ταπεινοφροσύνη. Έχει ανοίξει το δρόμο ο κύριος Φανρόμπα και είμαι βέβαιος ότι και με το Γενικό Γραμματέα του Λαϊκού Κόμματος σας υποστηρίζουμε όλοι μαζί σε αυτό το τεράστιο έργο που σας περιμένει. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Η κυρία Αντρικέων έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Συγχαίρω του συναδέλφους που συνέβαλαν τα μάλα στην πρόσπιση των θέσεων του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η... Για την δημιουργία αυτού του νέου σημαντικού θεσμικού οργάνου. Το αποτέλεσμα εξυπηρετεί και καλύπτει τα συμφέροντα και του Κοινοβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης εν γέννη. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να διατηρήσει την κοινοτική μέθοδο στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και την δυνατότητα ε, δημοσιονομικής παρακολούθησης. Είναι πολύ σημαντικό να επαναλαμβάνεται στο ψήφι που επαναλαμβάνεται στο ψήφισμα η γεωγραφική ισορροπία, κάτι που στη διαδικασία πρόσληψης των μελών της υπηρεσίας. Επίσης, η αρχή αυτή θα πρέπει να παραμείνει ισχυρή και να τηρείται και σε μεταγενέστερες φάσεις ε, της υπηρεσίας. Περιμένουμε πολλά από, την από τους επερχόμενους κανονισμούς προσωπικού και τον δημοσιονομικό κανονικό για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Άννα Γκόμες, ένα λεπτό. Εκτός μικροφώνου. Thank η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να οδηγήσει σε μια ευρωπαϊκή πολιτική αποτελεσματική και με νομιμότητα. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, όμως ε, λείπουν πολλά. Θα πρέπει να τηρήσουμε τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για ειρήνη και ασφάλεια που δεν ε, μπορούν να επιτευχθούν χωρίς ε, μια δημοκρατική διαδικασία και τήρηση των δικαιωμάτων των γυναικών. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα σωστά μέσα για να προωθήσουμε μια κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί παρά να τηρεί και τις ε, ε, προδιαγραφές που ορίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας των ε, Ηνωμένων Εθνών και θα πρέπει βεβαίως να τύχει αναθεώρησης και αυτό. Μιγκάλσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Χαίρομαι διότι επιτύχαμε μία συνένεση σε αυτό το σώμα ως προς το κριτήριο της γεωγραφικής εκπροσώπησης, διότι παρενέβη και το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές και η δική μου ομάδα. Ελπίζω τώρα να θεωρήσουμε τη σωστή γεωγραφική κατανομή ως κάτι δεδομένο. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δεν θα αντικαταστήσει τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι θα επικεντρωθεί σε αυτό που είπανε, πολύ προείπαν, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα ήθελα η ύπατη εκπρόσωπος να καταβάλει μια προσπάθεια έτσι ώστε πέρα από τη γεωγραφική κατανομή να ε, τηρηθούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ύπατη εκπρόσωπο ε, κανονικά πρέπει να πάρει εντολή από το Συμβούλιο, που περιλαμβάνει εκπροσώπου κρατών μελών. Ωστόσο, σήμερα ακούσαμε από του συζητητέ ότι η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να υπόκειται σε πανεθνικοποίηση, και ότι πρέπει να σπάσει τις κόκκινες γραμμές που θέτουν τα κράτη-μέλη. Ότι η εξωτερική πολιτική με λόγια πρέπει να είναι ελεύθερη από την παρέμβαση των κρατών μελών. Το Συμβούλιο πρέπει να δίνει εντολή στο συνήπατε εκπρόσωπο, αλλά τα μέλη του Συμβουλίου δεν πρέπει να παρεμβαίνουν. Η συζήτηση στην ΑΦΚΟ δείχνει σαφές ότι ε, το κοντινότερο όργανο στο οποίο θα είναι κοντά η υπηρεσία αυτή είναι η Κομισιόν, τη οποία η ύπατη εκπρόσωπο είναι και αντιπρόεδρο. Όταν ε, η συνθήκη τη Λισαβόνα αντικατέστησε τη συνταγματική συνθήκη, η Βρετανική κυβέρνηση περιέγραψε την ύπατη εκπρόσωπο ως απλό ε, και αυλαβή εκπρόσωπο των κρατών μελών για να μην υπάρξει κατηγορία ότι δημιουργείται ένα σούπερ υπερκράτος στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούχαν, τελευταίος ομιλητής, ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπαίνουμε σε, κάνουμε ένα βασικό και τελευταίο βήμα για τη δημιουργία της εξωτερικής υπηρεσίας ε, δράσης. Νομίζω ότι αυτό το βήμα θα πρέπει να ε, γίνει πολύ γρήγορα μέχρι το τέλος του έτους, έτσι ώστε να έχουμε και τις ε, τρεις πηγές που προβλέπει η συνθήκη για την πραγμάτωσή της. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη γεωγραφική κατανομή ως προς το προσωπικό στην ε, υπηρεσία αυτή. Τα νέα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα τα νεότερα κράτη-μέλη ε, όπως η Ρουμανία δεν έχουν σωστή εκπροσώπηση, έχουν αμεληταία εκπροσώπηση σε αυτή τη διάφρωση. Θα ήθελα να ρωτήσω την ύπατη εκπρόσωπο πώς μπορεί να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει σωστή θεώρηση του ζητήματος. Όταν μιλάμε δηλαδή για γεωγραφική κατανομή δεν είμαστε σαφείς ιδιαίτερα σε επίπεδο ε, διοίκησης. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας συνάδελφοι. Κύρια, ας τον έχετε το λόγο για να κάνετε παρατηρήσεις και να απαντήσετε στα ερωτήματα. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ και καταρχάς να ευχαριστήσω όλους όσοι εν γέννη μας υποστηρίξετε πλήρω ή εν μέρη. Όσοι δεν θεωρείτε ότι μπορείτε να υποστηρίξετε την πρόταση, ελπίζω να σα κερδίσουμε στο μέλλον και να καταλήξετε κι εσείς υπερήφανοι γι' αυτό που δημιουργήσαμε. Παρεπιπτόντως, εγώ ουδέποτε πρότεινα να έχω αεροπλάνο. Αν θέλετε να μου δώσετε, θα το δεχτώ, αλλά εγώ δεν το, δεν το ζήτησα. Να απαντήσω σε κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις ε, που ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι πολλές φορές. Κάτι που είπε η κυρία Λούνατσεκ. Να εξετάσουμε προσεκτικά την ισότητα ευκαιριών. Το θέμα δεν είναι μόνο ισότητα ευκαιριών αλλά και πρόσβαση να εξασφαλίσουμε ότι οι διαδικασίες που θεσπίζουμε επιτρέπουν και η γεωγραφική και η ισορροπία και παρουσία έμφυλη. Και θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία αυτή θα είναι ουσιαστική. Κάποιοι συνάδελφοί σας επίσης μίλησαν για τους πόρους. Καταλαβαίνω και αναγνωρίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε σωστά τους πόρους. Έχω απόλυτη επίγνωση ότι η οικονομική κατάσταση σήμερα είναι αυτή που είναι. Και διαφορετική ωστόσο να ήταν, θα ήθελα να έχω μια υπηρεσία που θα λειτουργεί σωστά και θα εκμεταλλεύεται με φιδό τους πόρους. Για το προσωπικό, επειδή πολλοί το ρώτησαν. Αυτή τη στιγμή έχουμε διπλωματικό προσωπικό 800 ατόμων, το 1 τρίτο των οποίων εκτός Ένωσης. Η Γαλλία, η Ισπανία έχει πάνω από χίλιους, η Γαλλία έχει 3.000, η Ολλανδία έχει 1.600 αντίστοιχους. Αυτό σας δείχνει μια εικόνα των διαστάσεων. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι ζητούμε από το προσωπικό να λειτουργεί στα πλαίσια της συνθήκης μετά την Λισαβόνα. Οι δουλειές που κάνουν δεν γίνονται πλέον από τα κράτη-μέλη, που σημαίνει ότι ορισμένε αντιπροσωπείε, η Νέα Υόρκη, η Γενέβη, θα πρέπει να καλύπτουν δραστηριότητες χωρίς άτομα. Εμείς λοιπόν θέλουμε να υπάρχει αποτελεσματική υπηρεσία ικανή να κάνει τη δουλειά της, τη δουλειά που εμείς συμφωνήσαμε να κάνει. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να υπάρχει διαφάνεια σε αυτό και θέλω να υπάρχει ε, ρόλος του Κοινοβουλίου και να ο ρόλος αυτός να διαδραματίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου και από την Επιτροπή Προπολογισμών. Στην ερώτηση του κύριου Λάμπστορφ, εγώ επαναλαμβάνω τη δήλωση που, έχω σήμερα, που έκανα σήμερα. Στο κείμενο της ε, συμφωνίας με το Κοινοβούλιο θα βρείτε αυτά που σας είπα και είναι σαφή κύριε Τάνοκ, θέσετε εκ νέου και εσείς και άλλοι ε, συνάδελφοί σας το θέμα της εμπλοκής των εθνικών κοινοβουλίων. Είναι κάτι ενδιαφέρον και οι δομές που θα θεσπίσω θα καλύπτουν και τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με τα εθνικά κοινοβούλια. Όταν πήγαινα μεταξύ Μόσχας, Κιέβου, Ισπανίας και Βρυξελών, όλο και στην Πάλμα, το έκανα μεταξύ άλλων διότι ήθελα να συναντήσω τους προέδρους των διαφορών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Εξωτερικών Υποθέσεων συγγνώμη, των κρατών μελών και θα το ξανακάνω και το φθινόπωρο στην συνάντηση που θα οργανώσει η Βελγική Προεδρία. Θέλω να ξέρω τι λένε τα, Ευρωπαϊ... τα Εθνικά Κοινοβούλια και προσπαθώ να βρω τον τρόπο για να ακούσω τι θα πούνε. Επίσης αναγνωρίζω ότι πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες για να μπουν νέοι, νέοι υπάλληλοι. Ε, υπάρχουν παραδείγματα όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την συνθήκη για να προσλάβουμε άτομα που έχουν την εμπειρογνωμοσύνη που θέλουμε. Κύριε Χάουταλ, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Θα συνεργαστούμε στενά με την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως ξέρετε, προσπαθώ να βελτιώσω τους στόχους μας και στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Κύριε Σάουριος Βόλτσκι, και σε άλλους το λέω αυτό, θέσατε το πολύ σημαντικό ζήτημα της γεωγραφικής εξισορρόπησης. Τι άλλο να σας πω. Εγώ δεσμεύομαι να το τηρήσω. Στην αναθεώρηση θα δείτε τι κάναμε. Αυτό που θεωρώ σαφές είναι ότι θα στηριζόμαστε θα, θα προσλαμβάνουμε αξιοκρατικά. Και μπορώ να σας πω ότι αυτό συμβαίνει ήδη γιατί έχουμε ξεκινήσει τις συνεντεύξεις. Άτομα που έρχονται από διαφορετικά τμήματα της Ένωσης. Ελπίζω σύντομα στην πρώτη αυτή ομάδα διορισμών και στην επόμενη που θα γίνει το Σεπτέμβριο και στην κεντρική δομή θα έχουμε και εξισορρόπηση γεωγραφική και εξισορρόπηση φύλου και αξιοκρατία. Βεβαίως για, το, για την εξισορρόπηση φύλου πρέπει να παροτρύνουμε την υποψηφιότητα περισσότερων και ό,τι κάνετε κι εσείς και εμείς τόσο το καλύτερο θα είναι στον τομέα αυτό. Για να επανέλθουμε στόσο στο θέμα της γεωγραφικής εξισορρόπησης και θα δείτε ότι θα το κρίνετε κι εσείς αλλά εγώ δεσμεύομαι απόλυτα. Σε ό,τι αφορά ο κ. Ντανζόν μίλησε για την ανάγκη να αυξηθεί η επιτόπη επίδοσή μας. Το κάνουμε νομίζω, το δείχνουμε. Ξέρετε ότι θα κάνω μια σειρά επισκέψεων τις επόμενες τρεις εβδομάδες την Μέση Ανατολή εκ όπου θα εξετάσω κατά πόσον η Ένωση θα έπρεπε να κάνει περισσότερα στην ε, περιοχή της, στη Λοίδα της Γάζας. Ξέρετε ότι ε, θα πάω στο Κυριστάν, έχει και μια συζήτηση σχετικά. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που προσπαθούμε να υλοποιήσουμε υποστηρίζοντας και τους ανθρώπους μας εκεί και τη δράση της Ένωσης, ιδίως στην ανθρωπιστική βοήθεια. Η κυρία Γεωργίευα κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί. Νομίζω ότι απάντησε στα μεγάλα ερωτήματα που τέθηκαν. Κλείνω όπως ξεκινώ. Ευχαριστώ πραγματικά όλους όσοι παρενέβησαν στη συζήτηση αυτή, τους συζητητές ιδίως, εσάς πρόεδρε, αλλά και τους βουλευτές που κουβέντιασαν μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι αυτό που δημιουργούμε τώρα είναι κάτι που πραγματικά θα σας κάνει Σας Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, είπατε πρόσωπε για τα σχόλιά σας. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξ ονόματος της Επιτροπής, κύριος Μάρος Χεύκοβιτς, έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε μεγάλη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νιώθω για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και πιστεύω ότι η αυριανή ψηφοφορία θα αποτελέσει ιστορικό ορόσημο για την Ευρώπη. Θα είναι η μέρα που η Ευρώπη θα βαδίσει προς ε, ισχυρότερη παγκόσμια ευρωπαϊκή παρουσία. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικεντρωθούμε όσο γίνεται περισσότερο στην ολοκλήρωση του έργου που απομένει μπροστά μας. Ε, απόφαση για τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, το δημοσιονομικό κανονισμό και ε, τον προπολογισμό. Όσο γίνεται καλύτερα. Είμαστε πρόθυμοι να διερευνήσουμε ε, όλες τις δυνατότητες όπου μπορούμε εμείς να παρέχουμε υπαλλήλου για την στελέχωση της υπηρεσίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν αυτό βοηθάει στο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα. Είμαι πεπισμένος ότι η ΕΕΔ θα μας φέρει περισσότερη συνεργασία, αποτελεσματικότητα, σαφήνεια, συνεκτικότητα και καλύτερες υπηρεσίες για τους Ευρωπαίους πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό και χρειάζονται ανάγκη και ε, έχουν ανάγκη υποστήριξη και βοήθειας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίφερ Χόφστατ, ε, εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που μίλησαν για την υποστήριξή του στον κύριο Μπρόκ, στον κύριο Γκαλτιέρη και σε μένα για τα αποτελέσματα που είχαμε στις διαπραγματεύσεις. Θέλω να πω μόνο ότι δεν καταλαβαίνω μερικές παρεμβάσεις εδώ μέσα που λένε όχι, όχι, όχι, τα έθνη, κράτη θα πρέπει αποκλειστικά να είναι αρμόδια για την εξωτερική πολιτική. Μα σε ποιον αιώνα ζείτε. Η τρομοκρατία σταματάει στα σύνορα, τίποτα. Των κρατών μελών, των εθνών. Ή μήπω η κλιματική αλλαγή. Πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει προβλήματα κλιματικής ε, ε, αλλαγής ότι όχι μόνο τα κράτη το συζητάνε και όχι η Ευρώπη. Μετανάστευση, Φερρυπίν, τα μεταναστευτικά ευρωπη μεταναστευση πιν τα μεταναστευτικα ρευματα διερωτώ πραγματικά. Έχω καμιά φορά την εντύπωση ότι πολλοί από τους συναδέρφους μας που είναι λίγο σκεπτικιστές ζουν ακόμα στο 19ο αιώνα, όπου τα έθνη κράτη αποφασίζαν τα πάντα με την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων στην Ευρώπη. Σε άλλο κόσμο ζούμε, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολυπολικό σήμερα ο κόσμος και η Ευρώπη είτε θα έχει λόγο ως Ευρώπη, είτε δεν θα έχουμε καθόλου φωνή. Ένα δεύτερο στοιχείο που λίγο με σοκάρει. θα κοστίσει χρήματα, λέει. θα κοστίσει το Το αντίθετο, κύριε Πρόεδρε, οικονομία θα κάνουμε με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Διότι για πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα να μειώσουν τις προξενικές τους υπηρεσίες σε πολλά κράτη του κόσμου. Είναι λοιπόν ένα εργαλείο εξοικονόμησης χρημάτων. Και από εκεί και πέρα είναι μια αρχή. Η υπηρεσία εξωτερική δράση είναι το διπλωματικό σώμα που χρειαζόμαστε για να έχουμε εξωτερική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέκαθεν πίστευα ότι πρώτα φτιάχνει διπλωματική υπηρεσία και μετά εξωτερική πολιτική. Χωρί αυτή την υπηρεσία δεν γίνεται. Αλλιώ προχωρούμε σε διαφορετικέ κατευθύνσει. Και ποιο είναι το επόμενο στάδιο, το γνωρίζουμε ήδη μεγαλύτερη συνεργασία για την ευρωπαϊκή άμυνα. Διότι ευρωπαϊκή διπλωματία χωρίς ευρωπαϊκή άμυνα, ε κάτι λείπει εκεί. Λοιπόν, προσεχώς ευρωπαϊκή άμυνα. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή άμυνα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σίγητα. Ο Έλμαρ Μπρόκ, άλλος εισηγητής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. 70% του πληθυσμού στην Ευρώπη σε όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο ποσοστό υπέρ της Ευρώπης από ότι σε αυτόν τον κλάδο. Και εκεί έχουμε την πιο ε, αδύναμη δράση. Οι λαοί το θέλουνε. Οι ελίτ δεν το θέλουνε στις πρωτεύουσε. Και έρχονται πάλι με την κυριαρχία αυτό που είπε ο κ. Σοφερχόφστατ, δεν κρεμίζουμε την κυριαρχία, τη συγκεντρώνουμε και την κερδίζουμε για τους πολίτες μας, γιατί έχουμε φωνή στον κόσμο και υπάρχουμε. Περί αυτού πρόκειται και τίποτα διαφορετικό. Και εκεί θα ε, συνεισφέρει η υπηρεσία αυτή. Κυρία Υπάτη, σας ευχαριστώ για τη δήλωση που κάνατε. Ε, θεωρώ ότι θα ενημερώνετε έτσι το Κοινοβούλιο και θα ε, δημοσιευτεί έτσι στην επίσημη εφημερίδα τα τυπικά θα τα ξαναπούμε, αλλά έχετε δεσμευτεί και τώρα ε, περνάμε στην εφαρμογή αυτής της προσπάθειας. Θα ήθελα επίσης να ξαναπώ ότι στη δίκαιη κατανομή των θέσεων και σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τις ε, πολύ ψηλέ θέσεις. Όχι μόνο οι πρόεδροι και οι γενικοί γραμματείς να είναι υπάλληλοι του Συμβουλίου, είναι στο εμπαρόδο και αυτό, και έχουμε και στο νομοθετικό ψήφισμα εκφράσει ορισμένα σχετικά. Το έχετε στα χέρια σας για τον κανονισμό υπηρεσιακή κατάστασης και διάφορα άλλα στοιχεία που θέλουμε ε, πέρα από τη συμφωνία. Λέει Άστον, θα ήθελα επίσης να σας πω το εξής. Βλέπετε εδώ ένα όγκο, μια στίβα χαρτιά που έχει μπροστά της η κυρία Γκρέστλε δεν είναι απειλή, αλλά αυξάνεται ήδη το ενδιαφέρον για την υπηρεσία σας από πλευράς Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κίφερ Χόφστατ και τον Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη για την πολύ καλή συνεργασία και σε ανθρώπινο επίπεδο πράγματι. Και όλους τους συναδέλφους, εσάς κυρία Υπάτη, ε, τον Πολ Κριστόφερσον και τους συναδέλφους Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιτρέψτε μου και πάλι τα εξαίρεση να ευχαριστήσω τους υπαλλήλου του Κοινοβουλίου, την κυρία Εύα Παλάτοβα που έκανε καταπληκτική δουλειά πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εκ νέου την κυρία Άστον για την λαμπρή δουλειά της και την συνεργασία με το Κοινοβούλιο τους τελευταίους μήνες. Ήταν πολύ σημαντικό για μας. Ευχαριστώ τους διαπραγματευτές μας, τον κύριο Σεύκοβιτς, τους συζητητές, τους επικεφαλείς των επιτροπών και την διαπραγματευτική ομάδα στο συνολό Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση τώρα.